Καλησπέρα σε όλους. Καροί κολέγοι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που προεδρεύω αυτή τη συνεδρίαση. Φυσικά ο πρόεδρος θα με αφήσει μόνο για λίγο. Αλλά καλό είναι και ένας αντιπρόεδρος να είναι χρήσιμος ε, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Έχουμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, η οποία έχει δύο αλλαγέ. Η πρώτη στο σημείο 5 για την τροποποίηση του κανονισμού 1098 του Βαλέσσα και μετά το πρωτόκολλο με την ε, Γουίνια Μπισάου προτείνεται να μεταφερθούν αύριο, για αύριο, να αναβληθούν για αύριο αυτά τα δύο σημεία. Το πρώτο ως πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης και το δεύτερο ως τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν είναι εδώ, ούτως ή άλλως θα ήταν αδύνατο να τα εξετάσουμε σήμερα αυτά τα θέματα. Ωραία, λοιπόν, εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Έτσι όπως παρουσιάζεται ανακοινώσεις της Προεδρίας υπάρχει μόνο μία σχετίζεται με την ε, προθεσμία τροπολογιών για την ΦΕΜ στη συνεδρίαση συντονιστών ορίστηκε ότι η προθεσμία θα είναι η 7η Δεκεμβρίου επόμενο Δεκεμβρίου για να ψηφιστεί στη συνέχεια βασική έκθεση ως τέταρτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε την παρουσίαση από τον Δ. Ρόμπερτ του, από το Πανεπιστήμιο του Ιόρκ το έγγραφο που αφορά τις ε, τοποθεσίες αποκαταστήσεις ε, θεμάτων. Γνωρίζετε ότι για αυτό το θέμα οι συζητήσεις που γίνεται στην Επιτροπή συχνά αξιολογούνται και περιλαμβάνονται και στη μεταρρύθμιση της ελληνικής πολιτικής. Πιστεύω ότι σήμερα αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να καταλάβουμε και το πόσο άξιζαν ορισμένα πράγματα που προτάθηκαν διαστητικά κιόλας από την Επιτροπή και που συζητήθηκαν εκτενώς. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα επιστημονικό έγγραφο το οποίο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα μας προσανατολίσει για τις συζητήσεις και για το τελικό έγγραφο του Κοινοβουλίου για την ε, κοινή ελευθερική πολιτική. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον ε, Δ. Ρόμπερτς, ο οποίος βρίσκεται εδώ και θα τον ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τα όσα θα μας ε, διηγηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη χαρά το να έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη στην ε, Επιτροπή Αλίας. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι για πολύ καιρό ερευνώ αυτό το τομέα ε, ε, μελετώ τα θαλάσσια καταφύγια που είναι ένα συνώνυμο των τοποθεσιών αποκατάστασης αποθεμάτων και αυτό αποτελεί ευκαιρία για μένα να σας ενημερώσω για τις γνώσεις που έχω αποκτήσει μετά από έρευνα δεκαετής ε, για αυτές τις τοποθεσίες. Η πρόταση, είχε γίνει πρόταση για μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής με προσθήκη μιας ε, τροπολογίας που θα λέει ότι οι τοποθέσεις αποκατάστασης αποθεμάτων θα πρέπει να οριστούν τέτοιες τοποθεσίες όπου θα απαγορεύεται οποιαδήποτε αλληλεία και αυτό θα επιτρέψει την αποκατάσταση των αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης ε, που υποβλήθηκε σε αυτή την Επιτροπή Αλίας, στην παρούσα Επιτροπή Αλίας, είναι ναι, η προοδευτική δημιουργία τοποθεσιών αποκατάσταση αποθεμάτων ε, στο 10 με 15% των εδαφικών χωρικών υδάτων έως 12 ναυτικά μελιά από τις ακτές. Εντός αυτών των τοποθεσιών αποκατάστασης θα απαγορεύεται οποιαδήποτε ελευτική δραστηριότητα και θα δημιουργηθούν αυτές οι περιοχές για την προστασία διαφορών οικοτόπων σημαντικών για εμπορικά ε, είδη ψαριών, όπως και ε, συμπεριλαμβανομένων επίσης και τόπων αναπαραγωγής ε, και οτοκίας των εχθείων. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ζώνων προστασίας γύρω από αυτές τις τοποθεσίες αποκατάστασης, όπου μόνο συγκεκριμένες ελευτικές δραστηριότητες θα επιτρέπονται. Αλευτικές δραστηριότητες με περιορισμένη χρήση εξοπλισμών, αλευτικών εξοπλισμών και χρήση γενικά εξοπλισμών με χαμηλές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Δηλαδή περισσότερο δίχτυα και καλάμια αντί για ε, τράτες βυθού, για παράδειγμα. Όπως είπα, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αποφασιστεί. Θα εξαπλωθεί σε μια σειρά ετών και Πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την επόμενη μεταρρύθμιση της, κοινής, της επόμενη μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής. Υπάρχει η δυνατότητα στο πλαίσιο της τροπολογίας να αλλάζει η τοποθεσία αυτών των περιοχών. Αλλά αρχικά τουλάχιστον η πρόταση λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για πέντε χρόνια, να οριστούν για πέντε χρόνια πριν αντικατασταθούν από άλλες. Πριν επιτραπεί να αντικατασταθούν από άλλες. Και φυσικά υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τη διέλευση αλευτικών σκαφών και υπάρχει μια ρήτρα μέσα στην προτινόμενη τροπολογία όπου λέει ότι τα αλευτικά σκάφη θα μπορούν να διέρχονται από αυτές τις περιοχές εφόσον έχουν αποθηκευμένο αλευτικό εξοπλισμό και αναγνωρίζεται ότι αυτές οι ε, περιοχές αποκατάστασης θα επηρεάσουν τη δομή στις τοπικές κοινότητες και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών κατά το χρόνο ορισμού αυτών των περιοχών αποκατάστασης. Αυτό που προτείνω λοιπόν να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα διαφορά στοιχεία που υπερασπίζουν τα πλεονεκτήματα σε αυτές, που προσφέρουν αυτές τις περιοχές αποκατάσταση στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε πόσο αποτελεσματικές έχουν υπάρξει στη διαχείριση της αλίας και να εξετάσουμε το εγκατάσταση των προστατευμένων περιοχών, θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών στην Ευρώπη και των καταφυγίων. Να κοιτάξουμε συγκεκριμένες διατάξεις της πρότασης σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, την κάλυψη αυτών των περιοχών και ούτω καθεξής. Αυτό που θα ήθελα να κάνω λοιπόν μέσα στα επόμενα 15 λεπτά είναι να σας παρουσιάσω τα κυριότερα ευρήματα αυτής της έκθεσης. Για να ξεκινήσουμε, για να καταλάβουμε την αξία και το ρόλο των περιοχών αποκατάστασης ηχθειαποθεμάτων στη διαχείριση της αλίας. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τον όρο Marine Reserve, σε θαλάσσια καταφύγια. Ο όρο τοποθεσίε αποκατάσταση ευθεία αποθεμάτων δημιουργήθηκε από αυτήν εδώ την Επιτροπή και ε, είναι συνώνυμο με αυτό που ονομάζουμε συνήθω τα επιστημονικά έγγραφα, θαλάσσια καταφύγια, marine reserve. Όταν αναφέρομαι λοιπόν σε θαλάσσια καταφύγια, ενώ τοποθεσίε αποκατάσταση ευθεία αποθεμάτων. Προτείναμε λοιπόν να προσφέρουμε ένα όφελο στην εμπορική αλία, επιτρέποντα την αποκατάσταση τη βιομάζα των ευθεία αποθεμάτων ώστε να αυξηθεί το μέγεθος οτοκίας για σημαντικά εμπορικά είδη μέσω εξάπλωσης που αποτελεί την καθαρή μετακίνηση των ζώων από το εσωτερικό μιας τοποθεσίας αποκατάστασης εκτός αυτής και στους, ε, στις αλληλευτικές τοποθεσίες για την εξαγωγή αυγών και προνεμφών, την παραγωγή νέων ζώων με την προστασία των πληθυσμών έτσι λοιπόν τα νεογνά μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης αυγών και προνυμφών από τις προστατευμένες περιοχές στα γύρω, στις τοποθεσίες. τα θαλάσσια καταφύγια μπορούν να προστατεύσουν ήδη εμπορικές σημασίες σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Ειδικότερα η πρόταση προτείνει προστασία κατά την οτοκία και κατά την φάση πολυνέρης ηλικία των ζώων. Ένας άλλο τομέας ε, επωφελής για τις αληθικές δραστηριότητες είναι η αποκατάσταση των οικοτόπων και η αυξημένη ποιότητα των οικοτόπων που προστατεύονται εντός αυτών των περιοχών. Τα ζώα έτσι μπορούν να ωφεληθούν από βελτιωμένες δυνατότητες, για παράδειγμα, ε, διατροφής. Τι στοιχεία έχουμε λοιπόν που υποστηρίζουν την αύξηση του μεγέθους ε, ότοκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα έχουμε πολύ ισχυρά ε, αξιόπιστα στοιχεία, πολλές ε, μελέτες έχουν γίνει μέσα στα χρόνια και αναθεωρήσεις και αυτή είναι μία από τις τελευταίες του 2009 και αυτό που βλέπετε είναι μία σειρά διαφορετικών μέτρων, μάλλον τρόπων μέτρησης των επιδόσεων αυτών των προστατευμένων περιοχών και εδώ βλέπετε ότι η γνωμάζα των ψαριών που αποτελεί το βάρος των προστατευόμενων ζώων αναμονάδα ε, οικοτόπου. Υπάρχει η πυκνότητα που είναι ο αριθμός ε, ζώων αναμονάδα ε, επιφανείας οικοτόπου και ο πλούτος που είναι ο αριθμός ειδών, το πλήθος ειδών προστατευόμενων ζώνων ανά μονάδα προστατευόμενης περιοχής οικότοπου. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε από αυτό το γράφημα είναι ότι τα θαλάσσια καταφύγια έχουν αυξήσει τη βιομάζα και την αυθονία και το μέγεθος και τον πλούτο των ειδών κατά μέσο όρο στις προστατευόμενες περιοχές σε σύγκριση με τις μη προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται κοντά ανάμεσα στο σημείο που βρίσκεται οι προστατευόμενοι, ε, τη, χρονική στιγμή προστασία τη περιοχή και κάποια άλλη στιγμή στον χρόνο. Έχουμε δηλαδή προστατευόμενε περιοχέ σε σύγκριση με μη προστατευόμενες και χρονική σύγκριση, δηλαδή πώ αλλάζει ο πληθυσμό από την εποχή ανάμεσα στο διάστημα προστασία και στο διάστημα στο οποίο έχει έρθει η προστασία. Το άλλο που πρέπει να εξετάσουμε είναι το ζήτημα του κατά πόσο αυτά τα θαλάσσια καταφύγια λειτουργούν σε εύκρατα νερά, όπως τα νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι όντω λειτουργούν, έχουν γίνει πολλέ μελέτε σε εύκρατε θαλάσσιε προστατευόμενε περιοχέ ε, όπω αυτέ και βλέπουν τις, ε, τα ίδια αποτελέσματα, ότι η προστασία παρέχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στις τροπικέ περιοχές. Ένα λοιπόν από τα επιχειρήματα που υπήρξε για χρόνια κατά του ορισμού των τοποθεσιών αποκατάσταση ε, ηχθιαποθεμάτων ήταν ότι δεν θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο σε εύκρατα νερά, το οποίο τελικά δεν συμβαίνει. Όσον αφορά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εξάπλωση, η εξάπλωση είναι η μετακίνηση των ζώων από μια προστατευόμενη περιοχή στα γύρω αλλιευτικέ περιοχέ όπου μπορούν να αλλιευτούν και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Έχει αποδειχθεί πολλέ φορέ ε, Έχουμε όλο και καλύτερα στοιχεία, αποκτούμε μια πιο ε, καλή εικόνα της αύξησης ε, της ποσότητας ε, ηχθείων και οστρακόδερμων που αλλιεύονται στις γύρω περιοχές, γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές σε πολλές περιπτώσεις. Στην Ευρώπη, ειδικότερα στη Μεσόγειο, υπάρχουν πολλά θαλάσσια καταφύγια δηλαδή τοποθεσίες αποκατάστασης, ε, όπου παρατηρείται εξάπλωση και η εξάπλωση μέσα στο χρόνο οδηγά σε συγκέντρωση της αλληλευτικής προσπάθειας κοντά στα σύνορα, στα όρια αυτών των θαλασσίων καταφυγίων και αυτό αποδεικνύει ότι συμβαίνει πράγματι η εξάπλωση και αυτά τα επιπλέον αλλιεύματα που βλέπουμε ε, ε, είναι πολύ κοντά στα όρια των θαλασσίων καταφυγίων. Έτσι μπορείτε να δείτε πώς οι ζώνες προστασίας, όπου επιτρέπεται μόνο συγκεκρι... επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες αλληλευτικές δραστηριότητες γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές και πώς αυτές οι περιοχές προστασίας είναι επωφελείς για ορισμένους τομείς ε, της αλίας. Αυτή η προσέγγιση έχει υιοθετηθεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, όπου ε, κοινότητες παραδοσιακής αλίας ε, λαμβάνουν πρόσβαση σε τέτοιες περιοχές κοντά στις προστατευόμενες περιοχές. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από το Κάμπο Τεπάλο στην Ισπανία, και όσο πιο ε, σκούρα είναι η σκίαση σε αυτό το γράφημα, τόσο πιο έντονη είναι η ελευτική προσπάθεια. Στην πάνω δεξιά πλευρά αυτής της εικόνας ε, βλέπετε μία λευκή κουκίδα και αυτή είναι η, περιοχή του θαλάσσιου κατηφυγίου όπου δεν επιτρέπεται αλία και βλέπετε πως οι αλληλευτικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται γύρω από αυτή την κουκίδα μία μακροπροθέσμη ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξάπλωσης ε, στη καταφύγια της Νότιας Ευρώπης ε, δείχνει αύξηση των αλλιευμάτων κατά 2 με 4% το έτος σε μεγάλο χρονικό διάστημα έως 30 χρόνια που είναι το μεγαλύτερο διάστημα που ληφθήκε υπόψη για μελέτη. Η άλλη πλευρά των ωφελών αυτών των θαλάσσιων καταφυγίων είναι η εξαγωγή νεογνών ζώων υπό τη μορφή ε, αυγών και προνεμφών. Τι συμβαίνει όταν προστατεύει κανείς ένα πληθυσμό, τα ζώα ζουν περισσότερα και γίνονται μεγαλύτερα ως ενηλικά ζώα, διότι η ποσότητα ε, νεογνών αυξάνεται γεωμετρικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, υπάρχει τεράστια, παρατηρείται τεράστια αύξηση αριθμού νεογνών και βλέπουμε τεράστιες αυξήσεις αναπαραγωγής ε, στον προστατευόμενο πληθυσμό σε αυτά τα θαλάσσια καταφύγια. Αυτός ο πληθυσμός μεταφέρεται στα γύρω, στις περιοχές και αυτή η εξαγωγή των αυγών και των προνυμφών στις γυροληφτικές περιοχές έρχεται από διάφορες πηγές ε, Κάναμε μελέτης για τις γενετικές ομοιότητες των πληθυσμών κατά μήκος παράκτων περιοχών για να δούμε πόσο μακριά πηγαίνουν, μετακινούνται τα νέα ζώα. Κάναμε οκεωνογραφικές μελέτες ε, με ε, μελετώντας τα ρεύματα και τις κατευθύνσεις των ρευμάτων ώστε να ε, διαπιστώσουμε πώς μετακινούνται αυτά τα νέα ζώα. Και έτσι λοιπόν η εξάπλωση αυγών και προνυμφών διαπιστώθηκε ότι μπορεί να καλύψει από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιόμετρα. Όταν έχουμε λοιπόν μια τοποθεσία αποκατάσταση ηχθεία αποθεμάτων, αυτή μπορεί να παρέχει αυγά και προνύμφες σε πολύ μεγάλη περιοχή γύρω από αυτήν. Αυτό που είδαμε ειδικότερα σε κάποιες ε, ειδικέ μελέτες πρόσφατες ε, συνέδεσαν ουσιαστικά απευθεία τα γονικά ψάρια πούμε, που αναπτύσσονταν μέσα στι προστατευόμενε περιοχέ με τα νεονά του που βρέθηκαν εκτό. Και η σημαντικότερη μελέτη έγινε στο Great Barrier Reef, δημοσιεύτηκε φέτο στην Αυστραλία και ε, διαπιστώνει μια βασική αρχή ε, που διέπει τη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών ε, ως υποστήριξη της διαχείρισης της αλίας είναι ότι ο πολλαπλησιασμό του πληθυσμού είναι αναλογικός με το ποσό αποθέματος που προστατεύεται εντό της προστατευόμενης περιοχής. Αυτό ακριβώς ε, ε, διαπιστώθηκε στο Great Barrier Reef στην Αυστραλία. Μία από τις πιο λεπτομερείς μελέτες που έγινε όσον αφορά τις διαπιστώσεις για την αλληλεία των θαλασσιών καταφύγιων στην Ευρώπη έγινε στα νησιά Κολουμπρέτες ε, και στο σχετικό θαλασσιό καταφύγιο στην Ισπανία. Εκεί προστατεύεται ένα αστάκου και Η μελέτη εξέτασε 5.000 αστακούς εντός της προστατευόμενης περιοχής και έδειξε ότι περίπου 4,7 των αστακών ε, 100 ε, των αστακών έφυγαν από την προστατευόμενη περιοχή εντός ε, του έτους ήταν πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος από αυτούς που υπήρχαν μέσα στο καταφύγιο και αποτέλεσαν σημαντικό ποσοστό των συνολικών αλλιευμάτων στις γεροαλλιευτικές περιοχές. Ε, ε, σχεδόν 31 με 43% των συνολικών αλλιευμάτων φυσικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη η συρρήκνωση των αλλιευτικών περιοχών που προκύπτει, αλλά παρόλα αυτά τα αλλιεύματα είναι κατά 10% υψηλότερα ως αποτέλεσμα της ύπαρξης της προστασίας αυτής σε αυτό το θαλάσσιο καταφύγιο. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι ο προστατευόμενος πληθυσμός συμβάλλει κατά 80% των αυγών που εμπλουτίζουν τον πληθυσμό ε, στην περιοχή επειδή έχουμε 80% μεγαλύτερη αναπαραγωγή εντός της προστατευόμενης περιοχής. Έτσι λοιπόν μπορεί να δει κανεί πώς τα πλεονεκτήματα της προστασίας ε, επηρεάζουν πολύ μεγαλύτερες περιοχές ε, τριγύρω. Φυσικά αυτό που συχνά ρωτάει είναι ορισμένοι όσον αφορά το πώ τα είδη υψηλή κοινωτικότητα επωφελούνται από αυτή την ύπαρξη αυτών των περιοχών, των προστατευόμενων περιοχών. Λένε λοιπόν ότι στα ευρωπαϊκά ύδατα δεν αναμενόταν ότι θα ήταν υποφελεί αυτέ οι περιοχέ, επειδή τα είδη κινούνται πάρα πολύ, συνεπώ δεν μπορεί να προστατεύονται επαρκώ μέσα σε αυτές τι συγκεκριμένες περιοχές. Στην πραγματικότητα όμω υποφελούνται με πολλού τρόπου και ήδη χρησιμοποιούμε προστατευόμενε περιοχέ ε, ε, ενό πιο περιορισμένου τύπου για να προωθήσουμε τις περιοχές οτοκίας ε, για κάποια συγκεκριμένα είδη και τη βιομάζα επίσης ε, αναπαραγωγής ε, και όπως είπαν νωρίτερα το είδος των οικοτόπων, το μέγεθος των πηγών ε, διατροφής στις προστατευόμενες περιοχές μπορεί επίσης να υποφελήσει και τα είδη υψηλής κινητικότητας καθώς μετακινούνται. Πώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι αυτά τα είδη υψηλής κινητικότητας υποφελούνται. Βάσει μιας ανάσης υπόθηκε ότι αυτά τα είδη ανα αποκρίθηκαν στην προστασία στα ε, θαλάσσια καταφύγια στην Ευρώπη και είπαν ότι αυτό ήταν ένα από τα εντυπωσιακότερα ευρήματα ότι τα είδη υψηλή κινητικότητα υποφελούνται ανεξαρτήτως της μετακίνησής τους. Ενώ θα θεωρούσε κανείς ότι θα συνέβαινε το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική έκθεση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, που έχει συμπεριληφθεί παλιότερα σε μια κοινοβουλευτική έκθεση εδώ του εδώ Κοινοβουλίου είναι η, περίπτωση του μπακαλιάρου στο της στη Σουηδία. Σε αυτά τα στενά δεν χρησιμοποιούνται ε, κινητή αλλιευτική εξοπλισμό από τη δεκαετία του 90. Χρησιμοποιούνται δίκτυα και ε, ε, καλάμια. Και αυτό που συνέβη είναι ότι η περιοχή στο κάτεγκατο που χρησιμοποιούνταν ε, γρηγροί ε, και τράτες ε, παρουσίασαν μείωση των αποθεμάτων ενώ στο Ωρεσούντ αυτά τα αποθέματα δεν μειώθηκαν και αν δούμε τη διαφορά πυκνότητας θα παρατηρήσουμε ότι η αυθονία είναι 40-50 φορές μεγαλύτερη στο Ωρεσούντ και αν δείτε τις φωτογραφίες ε, των μπακαλιάρων σε αυτή την προστατευόμενη περιοχή, είναι μεγάλα ψάρια, πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος από ό,τι βρίσκει κανείς σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα μιας μερικώς προστατευόμενης περιοχής, δεν είναι καν πλήρως προστατευμένη, ε, που υπήρξε ιδιαίτερα υποφελής ε, ως διαδικασία για, την, για τα συχθείες. Με ένα άλλο έβριμα αυτής της έκθεσης σχετίστηκε με το χρόνο απόδοσης των ωφελών για αυτά τα εχθή αποθέματα. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει, να εντοπίσει τα αποτελέσματα για τους προστατευόμενους πληθυσμούς εντός ήδη ενός-δύο έτων μετά από την έναρξη της προστασίας και μετά αυτό αυξάνεται αρκετά γρήγορα με το χρόνο εντός 5-10 ετών μετά από την έναρξη της προστασίας βλέπει κανείς σημαντικά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα και για την αλληλεία. Και το, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα ωφέλη συνεχίζουν να αυξάνονται για δεκαετίες μετά. Οπουδήποτε είχαμε μακροπρόθεσμες μελέτες αποθεμάτων, βλέπουμε ότι τα, τα ωφέλη αυτά αυξάνονται γεωμετρικά και συσσωρεύονται με τα χρόνια. Ε, σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρούμε ε, να σταματάει αυτή η αύξηση σε κάποιο ψηλό επίπεδο με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που είχαμε και για την αλία με την προστασία ε, αυτή ήταν πολύ πιο, ε, πιο σημαντικά τα αποτελέσματα από ό,τι νομίζαμε. Πόσο λοιπόν πρέπει να τώρα προστατεύουμε σύμφωνα με την πρόταση 10 με 20% των ε, υδάτων και αυτά εξαπλώνοντας το 20 με 30% της θάλασσας και σίγουρα είναι χρήσιμο να έχουμε ίσως το ανώτερο ποσοστό που προτείνεται εδώ των ε, ε, εθνικών υδάτων στο 20%. Πόση τέτοια προστασία έχουμε στην Ευρώπη ήδη. Κοιτώντας τα θαλάσσια καταφύγια στην Ευρώπη, οι καταστάσεις ε, είναι πολύ διαφορετικές ε, βλέπετε τη θάλασσα περιοχή ΟΣΠΑΡ στα αριστερά και τη Μεσόγειο θάλασσα στα δεξιά. Γενικά η εικόνα μοιάζει και στις δύο περιοχές. Έχουμε πολλές προστατευόμενες περιοχές, αλλά δεν καλύπτουν πολύ μεγάλο κομμάτι της θάλασσας. Και αν σκεφτεί κανεί πόσο ακριβώς, πόσο ακριβώς είναι η περιοχή της θάλασσας που προστατεύεται σε σχέση με το προτινόμενο ποσοστό, είναι ουσιαστικά μόλις το 1-16 χιλιοστό της περιοχής. Ε, ενώ ουσιαστικά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείτε αυτό το ποσοστό του 10-20% για την προστασία των περιοχών. Ορισμένα κρατημέλη έχουν ήδη εκτενή δίκτυα προστασίας ε, συγκεκριμένων περιοχών, αλλά η προστασία είναι γενικώ σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτή που προτείνεται. Θα υπήρχε ωστόσο η δυνατότητα, δεδομένη τη προσπάθεια που έχει επενδυθεί για τον ορισμό αυτών των περιοχών και για τι διαβουλεύσει με τι τοπικέ κοινότητε, να μετατραπούν σε τοποθεσίε αποκαταστάσει εχθεί αποθεμάτων, αναβαθμίζοντα το επίπεδο προστασία εντό αυτών των περιοχών. Από εμπειρία από άλλα μέρη του κόσμου παρατηρείται ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό με τη βοήθεια της αλληλευτικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία της και η στήριξή της ε, δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί για τη δημιουργία περιοχών προστασίας. Αυτή ήταν η εμπειρία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά στις περιπτώσεις όπου η βιομηχανία συμμετείχε στη διαδικασία από την αρχή με ουσιαστικό τρόπο τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά τα δίκτυα προστατευόμενων περιοχών υψηλής ποιότητας ε, που προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας ε, ε, δημιουργήθηκαν τέτοια δίκτυα επιτυχώς σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα κυρία βρήματα και συστάσεις από την έκθεση. 10 με 20% των χωρικών υδάτων θα βοηθούσαν να παρασχεθούν σημαντικά ωφέλη για τη βελτίωση των αποθεμάτων και την προστασία των οικοτόπων θα ήθελα να, να πω ότι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις για την προστασία και για τη διαχείριση της αλληλείας. Ε, είναι η σημαντικότερη πρόταση από όσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Θα ήταν τόσο απαραίτητο να υπάρχουν τέτοιες υψηλά προστατευόμενες περιοχές ώστε να βελτιώσουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβάλλον στο πλαίσιο της οδηγίας θαλάσσιας στρατηγικής όπου γίνεται έκκληση για ύπαρξη χρήση τέτοιων περιοχών προστατευόμενων ως εργαλείου για τη βελτίωση της κατάστασης των θαλασσών. Αλλά ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας ώστε να διατηρηθεί αυτό το υψηλό επίπεδο του θαλάσσιου περιβάλλοντος ορισμό λοιπόν τέτοιων περιοχών σε ποσοστό έω 20% των αλλιευτικών περιοχών και, στα χωρικά, και των χωρικών υδάτων θα μπορούσε να αυξήσει το όφελος που θα αποκομίσουμε από αυτές τι προστατευόμενες περιοχέ. Έτσι θα προωθηθούν τα συμφέροντα των αλλιέων μικρή κλίμακα και παραδοσιακών αλλιέων που λειτουργούν σε εθνικά ύδατα με μικρά σκάφη, όπου συμβαίνει συνήθω στην Μεσόγειο θάλασσα. Κάτι σημαντικό πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι αυτή δεν είναι μια πολιτική όπου απλά μπορούμε να πούμε θα το κάνουμε για πέντε χρόνια και μετά όλα θα είναι εντάξει και μετά μπορούμε να ξαναψαρεύουμε οπουδήποτε. Ουσιαστικά τα ωφέλη συσσωρεύονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλά μπορούν να καταστραφούν πάρα πολύ γρήγορα εφόσον ξαναξεκινήσει η αλία και αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ουσιαστικά ότι αν ξανανοίξουμε μια προστατευόμενη περιοχή ε, εξαλείφουμε όλα αυτά τα ωφέλη ε, όσον αφορά την αποκατάσταση αποθεμάτων για να λειτουργούν αποτελεσματικά αυτές οι περιοχές πρέπει να συμμετέχει και η αλληλευτική βιομηχανία. Η βιομηχανία της αλίας ουσιαστικά μπορεί να αποφασίσει για την υλοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου διαχείρισης ε, των αλληλευμάτων Δεδομένου του πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό και δεδομένου τη ανάγκη ευαισθητοποίηση στι ε, περιφερειακέ διαφορέ και στο περιβάλλον και στι κοινωνικέ συνθήκε, ε, σκόπιμο θα ήταν να εμπλέξουμε τα περιφερειακά ε, τις περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές για την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι θα είναι κάτι ακριβό, αλλά θα είναι αποτελεσματικό ω προ το κόστο μέσα στο χρόνο. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε διάφορε περιοχέ του κόσμου. Η δημιουργία λοιπόν τέτοιων περιοχών θα αποτελέσει επένδυση για το μέλλον. Αλλά θα υπάρχουν μεταβατικά κόστη. Αυτά τα μεταβατικά κόστη, εάν, εάν δεν επενδυθούν αυτά τα μεταβατικά κόστη, η επιτυχία δεν είναι τόσο διασφαλισμένη ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το θαλάσσια ταμεία ώστε να μπορέσουμε να να κάνουμε αποτελεσματική αυτή την πρόταση. Ε, επίσης, τα σκάφη, όπως είπαμε, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται να διέρχονται μέσα από αυτέ τι περιοχέ, απλά θα πρέπει να ε, διέρχονται με, ε, έχοντας, πληρώντας κάποιες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λυπάμαι γιατί έφτασα αργά. Έπρεπε να λάβω το λόγο σε μια άλλη επιτροπή, αλλά επανήλθα. Η κυρία Φράγκα ζήτησε το λόγο πρώτα απ' όλα, εκ μέρους των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ομιλητή για την ε, έκθεσή του. Εγώ είμαι Ισπανίδα, είμαι από μια χώρα στην οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραδοσιακά υπάρχουν αυτά τα θαλάσσια καταφύγια και συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο με εξαιρετικά αποτελέσματα, αποτελέσματα τουλάχιστον στη χώρα μου και έχει μειονεκτήματα διότι ο έλεγχος είναι δαπανηρός διότι το θέμα δεν είναι να κάνουμε αυτό το καταφύγιο, πρέπει να κάνουμε και διεξοδικού ελέγχου. Αλλά η συντήρηση είναι δαπανηρή. Βάση περιπτώσει, είναι αυτή η οικονομική διάσταση που σε εποχή οικονομική κρίση είναι σημαντικό. Τώρα, αυτά τα θαλάσσια καταφύγια, την άποψή μου, πρέπει να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον που θα έχουμε μία ενοποιημένη πολιτική αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το όλο σύστημα. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε στην αλληλεία όπως εσείς, θα πρέπει να το συνδυάσουμε και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι μιλούμε για επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέσο το οποίο θα πρέπει, όπως είπα, να διαδραματίσει το μέλλον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βασικά, βασικά όσον αφορά και τη διάσταση του οικοσυνείδηματος, διότι αν δεν έχουμε αλληλεία θα έχουμε άλλου τύπου ε, επιπτώσεις, την αιωλική ενέργεια και τις συνέπειες και άλλες δραστηριότητες οι οποίες απορρέουν. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει το οικοσύστημα να το δούμε σφαιρικά. Γι' αυτό μιλώ επίσης ότι έχουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον τα θαλάσσια καταφύγια. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μιλούμε και πάλι μόνο για την αλληλεία, για, αλλά γενικότερα για το οικοσύστημα και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες επιτροπές όπου είναι αυτό το οικοσύστημα το πιο ευαίσθητο. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να πω ότι το να μιλούμε για ποσοστά όπως γίνεται στην πρόταση της Επιτροπής και ειλικρινά και εσείς στην πρότασή σας νομίζω ότι μπορούν να είναι μια πάρα πολύ καλή προσδοκία αλλά δεν είναι εφαρμόσιμο στην πράξη. Διότι τελικά σε κάποιο μέρο χρειάζονται περισσότερα καταφύγια, σε λιγότερα. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα η Ιρλανδία, όπου μιλούμε για 30% ε, και για τη Μάλτα με το ίδιο ποσοστό του 30%. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα ποσοστά, να πούμε καλύτερα, ότι θα μπορέσουμε εκεί που είναι απαραίτητο να τα καθορίσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να καθορίσουμε εκ των προτέρων ε, ποσοστά. Δεν έχουν λογική για μένα. Είπα ότι θα πρέπει, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να τα έχουμε, να τα καθορίσουμε ένα ποσοστό που θα εξαρτάται από τη χώρα, από τη ζώνη, από τη θάλασσα κτλ. Αυτά ήταν τα σχόλια που ήθελα να κάνω βασικά όσον αφορά αυτή την διάσταση, την οικοσυστημική, την οποία νομίζω ότι έχετε κάπως παραγνωρίσει, αλλά επαναλαμβάνω το λέω αυτό για το μέλλον της αλίας. Ευχαριστώ κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Φράγκα. Με πλήσουν οι τελευταίοι αριθμοί, αλλά ο αριθμός αυτών των καταφυγιών υπάρχουν. Τι είπατε στην ε, Μεσόγειο, εν δέκατο του 1%. Καλά κατάλαβα. Χίλια. Ε, yeah, I mean... Τώρα, το κόστος. Νομίζω ότι είναι στην πράξη θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τους ενδιασμούς και την αντίσταση εκ μέρους των αλλιέων. Πώς μπορούμε να έχουμε την υποστήριξή τους και με τι κόστος, με πόσο κόστος. Τι σημαίνει αυτό. Συνειδητοποιώ ότι έχουμε και τις τροπολογίες του MMF που θα έρθουν ως ο νούπο, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε και ίσως είναι τώρα και τα Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ερευνητή για την έκθεση του. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές. Παντού στην Ευρώπη οι αλλοί σήμερα αγωνίζονται να συνεχίσουν να έχουν μία υφόρο δραστηριότητα έχουν να κάνουν με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, με την ε, μείωση των ε, ηχθειοποθεμάτων και θέλουν η δουλειά τους να αποδίδει για να μπορούν να ζουν από αυτήν. Η πρόταση αυτή, όπως μας δείχνουν οι επιστήμονες, μπορούν να αναστρέψουν αυτή την τάση, δηλαδή να αυξήσουν τα αποθέματα για τους αλληλείς, να κάνουν ε, σωστά οικοσυστήματα και οι υγιείς κοινότητες οι οποίες θα ασχολούνται με το επάγγελμα με το οποίο ασχολήθηκαν για χρόνια. Και μας δείχνει πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα αποθέματα αλλιευμάτων, να προστατεύσουμε τις θάλασσες και τους αλλιήμνες μας βεβαίως. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο 20%. Είδα αυτό της στάσεις και το Κοινοβούλιο προτείνει τα μέτρα και οι προτάσεις αυτές να γίνουν με την συμμετοχή των ενεχομένων. Να αποφασιστούν από τις τοπικές κοινότητες, από τους επιστήμονες, από τους επαγγελματίες του κράτους αλληλής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι δυνατόν. Έχει συμβεί ήδη σε πολλές περιοχές όπου ολοκληρώθηκε αυτή η πρόταση και εφαρμόστηκε. Και κατανοούμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος για την αναγέννηση των νυχθειοποθεμάτων στην Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αλληλείς μας ώστε να αλλιεύουν μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά συγχρόνως να αποκαθίστανται και να αποθένται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας, όχι κυρία Τόμας, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρόμπερτς Συμμερίζομαι και εγώ την ιδέα ότι τα αποθέματα είναι πολύ σημαντικά. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα γενικότερα. συμπεραίνετε και επιμένετε ότι θα πρέπει αφενός να έχουμε κλείσιμο σε ποσοστό 20% και απ' την άλλη λέτε ότι κάποια στιγμή, το είπατε στην έκθεσή σας, εάν ξανανοίξουν αυτές οι ζώνες θα χάσουμε όλα τα ωφέλη. Όταν όμως χρησιμοποιείτε παραδείγματα και το καλύτερο είναι αυτό του γάδου, έχουμε να κάνουμε με μία μερική ζώνη. Τώρα, μπορούμε να βρούμε και άλλες ζώνες, τις οποίες η αλία είναι εποχική. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, δεν θα πρέπει το είδος του καταφυγίου να είναι προσαρμοσμένο στα είδη, στα οικοσυστήματα και στους στόχους τους οποίους θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον Κρήτον Αρσένη ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο τοπική προσέγγιση με τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες του κλάδου. Δεύτερο ερώτημα που μου δημιούργησε απορίες περιγράφεται στην Ισπανία κάποια ζώνη και λέτε αν σας κατάλαβα καλά ή δεν είμαι και σίγουρη ότι ετησίως παρατηρείται 2 με 4 αύξηση στις ε, περιφερικές ζώνες της ζώνης, που περιγράφεται αλλά αν πρόκειται για περιοχές γύρω από την προστατευόμενη ζώνη ποσοστού 2-4% τα ωφέλη είναι τόσο μεγάλα όσο λέγεται. Απ' την άλλη, εάν λέτε αύξηση 2 4% ετησίως, η έκθεση έγινε με εγγύς ζώνες συγκρίσιμες για να μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα πιο σφαιρική. Και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Φράγκα προηγουμένως για το γεγονός ότι όντες οι ζώνες αποκατάστασης στην αλληλεία ε, είναι κάτι το θετικό, αλλά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται και άρα δεν μπορούμε αποκλειστικά να μιλούμε για αλληλεία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή. Πολλά έχουν ήδη υποθεί, γι' αυτό θα περιοριστώ σε ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις που έχω προσωπικά. Είπατε στην παρουσίασή σας ότι εν μέρει προστατευόμενες περιοχές ε, μπορούν επίσης να έχουν επιτυχία. Μπορείτε να το ορίσετε επακριβώς τι σημαίνει μερικώς προστατευόμενες περιοχές και ποιο θα πρέπει να είναι το μέγεθός τους. Επίσης με ενδιαφέρει το εξή να μας πείτε το εξή. Είπατε ότι η αληφτική βιομηχανία θα πρέπει να αποφασίσει να κρίνει πού θα πρέπει να, ε, πού θα πρέπει να τοποθετούν αυτές οι προστατευόμενες περιοχές. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στην μετάφραση ε, ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η αλευτική βιομηχανία είναι σε θέση να κρίνει, να αξιολογήσει πού θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτές οι περιοχές. Θεωρώ ότι είναι πολιτικό ζήτημα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες και αν θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια ποσοστά, τι σημαίνει σε χώρες που έχουν μικρή ακτογραμμή, για παράδειγμα στο Βέλγιο μπορούμε να πετήσουμε από το Βέλγιο αυτό το ποσοστό του 20% γιατί τότε καλύπτεται ολόκληρη η ακτή του Βελγίου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλω να με παρανοήσετε, αλλά θα ήθελα πραγματικά να το κάνουμε ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Πιστεύω ότι λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα. Και σημαντικό είναι, όπως είπε ο Κρις και η κυρία Φράγκα, ότι όλα αυτά συνεπάγονται ένα κόστος. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια οικονομική υποστήριξη. Για σκεφτείτε να κάνετε μια έρευνα επί 20 χρόνια. Θα έχετε μια αντίληψη ε, που κινείται το κόστος αυτής της χρηματοδοτικής υποστήριξης, ενίσχυσης. Θα ήθελα να μας πείτε κάποιους αριθμούς από το ελάχιστο έως το μέγιστο ποσό, γιατί θεωρώ τέτοια νούμερα θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικά. Ο κύριος Ρωμέρο έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, πιστεύω ότι το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι το γεγονός ότι μας εξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ζώνες το θέμα είναι, το πιο σημαντικό είναι το πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι και το ζήτημα της πολιτικής. Πολλοί συμφωνούν για το γιατί, αλλά όλοι δεν συμφωνούν για το πώς πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει σχετική συζήτηση. Ε, αλλά αν πάρουμε κάποια παραδείγματα και πήρα, αναφέρατε κάποιο παράδειγμα στην Ισπανία ή κάποιες άλλες χώρες, έχετε κάποιες σχετικές εμπειρίες όπου η αλία μικρής κλίμακας οι ίδιοι ελείς προωθούν τέτοιου είδους ε, προστατευόμενες περιοχές ή θαλάσσια ε, καταφύγια. Υπάρχει μια κατανόηση εκ μέρους του κλάδου. Άρα υπάρχει μια κατανόηση εκ μέρους του κλάδου που θεωρούν ότι είναι ωφέλιμο για αυτούς να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται για μια περιχαράκωση, ένα κλείσιμο κάποιων περιοχών, αλλά ένα τρόπο τελικά ε, μελλοντικής επένδυσης ε, στο θαλάσσιο πλούτο, στα θαλάσσια αποθέματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ότι όταν δεν μιλούμε μόνο για πολιτική βούληση, αλλά και για δημόσιες επενδύσεις, είναι σημαντικό να μπορούμε να πείσουμε όλους όσους επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις, πολίτες. Ε, αναφέρθηκε το MMF, νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακεί εδώ και θα πρέπει να εξηγήσουμε επίσης ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα κόστους αυτού του θαλάσσιου καταφυγίου, το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί, αλλά τα πλεονεκτήματα τα οποία θα παραχθούν θα είναι σημαντικά και δεν θα υπάρξουν αν δεν γίνει με ένα σωστό τρόπο. Εάν εστιάσουμε μόνο στο κόστος, της, αυτών των θαλάσσιων καταφυγίων, των προστατών περιοχών, νομίζω ότι δεν θα πείσουμε απολύτω κανένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιλάνα. Όπως γνωρίζετε όλοι, εγώ έχω πιστεί για αυτό το ζήτημα. Το έχω συζητήσει πολλές φορές, κατά επανάληψη. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη πράξη που θα μας βοηθήσει να μετασχηματίσουμε την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική, δίνοντάς της μια δυνατότητα χωροταξίας της θάλασσας. Πιστεύω ότι δεν είναι το παν. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ελευτικές δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρούν τη θάλασσα μόνο ένα μέρος όπου αλλιεύουν και όχι χώρος όπου καλλιεργούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να υποστηρίξουμε μια τέτοια θέση παρέχοντας τους πόρους. Εγώ θέλω να προτείνω τρία απλά πράγματα. Εμείς σήμερα με τις ε, ε ουσιώδεις παρεμβάσεις χρηματοδοτούμε χρόνο μη Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε χώρο μη μειώνοντας σταδιακά το χρόνο μια αλληλίας που χρηματοδοτούμε και αυξάνοντας το χώρο. Χωρίς να κάνουμε καμιά τεράστια επανάσταση, αλλά ώστε βαθμία αυτό να αποτελέσει μια πολιτική που θα παρέχει προοπτική. Δεύτερο στοιχείο. Πώς θα το αποφασίσουμε. Εμείς συμμετέχουμε σε μια επιτροπή όπου το σημαντικότερο βάρος της οικονομικής δραστηριότητας σήμερα στην Ευρώπη εκπροσωπείται από τους αλληλείς. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μαζί με τους αλληλείς. Ναι, με τους επιστήμονες, ναι και με τα κρατημέλη, αλλά και με τους αλληλείς. Πραγματικές συμφωνίες που να βασίζονται στην στο χωραταξικό σχεδιασμό. Τρίτο στοιχείο, ο έλεγχος. Σήμερα ο έλεγχος των καταφυγίων, των περιοχών αυτών είναι δύσκολος. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν οριστεί με ακρίβεια. Μερικές φορές βρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα, άλλες φορές αλλού. Αλλά όπως αναφέρουμε στην τροπολογία 68-0,12 μίλια για από την ακτή σημαίνει ότι οποιοδήποτε σκάφος μπαίνει σε αυτό το χώρο θα μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Η ιδέα αυτή λοιπόν απλούστευση των ελέγχων είναι θεμελιώδη σημασία. Τελευταίο ζήτημα που ήθελα να αναφέρω, εάν δεν υιοθετήσουμε αυτή την επιλογή, εμείς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το MSY, με, το, με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εάν δεν υιοθετήσουμε μια επιλογή βάσει της οποίας η θάλασσα θα παράγει περισσότερα, οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές για τον τομέα της ελίας. Διότι η, εφαρμογή, η ε, μη εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα δημιουργήσει φρικτά αποτελέσματα για τον τομέα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Μερικοί λένε μέχρι το 2015, μέχρι το 2016. Θα έχει φοβερά αποτελέσματα. Θα οδηγήσει στο θάνατο του τομέα. Αυτό το 0,001% που αναφέρθηκε και λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Δέβης, φαίνεται πολύ δύσκολο να περάσουμε από το 0,01% στο 20%. Μπορεί να φαίνεται τεράστιο άλμα. Εγώ πιστεύω ότι στο 0,01% βρίσκονται μόνο οι καθορισμένοι προστατευμένοι χώροι. Αλλά οι περιοχές όπου δεν ε, υπάρχουν αλληλευτικές δραστηριότητες είναι περισσότερες. Εγώ πιστεύω ότι υπολογίζοντας αυτό το 20% θα πρέπει να υπολογίσουμε και όλες τις υπόλοιπες αλληλευτικές ε, δραστηριότητες, τους χώρους που έχουν αφιερωθεί στις εκθεοκαλλιέργειες... Για παράδειγμα, έτσι λοιπόν πιστεύω εγώ σήμερα, ε, πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα ποσοστά το οποίο είναι περισσότερο από το 5-6%. Το να περάσουμε λοιπόν από το 5-6% στο 10% στο 20% εντός 10 ετών δεν είναι τόσο αδύνατο. Ξεκινώντας όμως με φετρία την ιδέα ότι σήμερα προστατεύεται μόνο το 0,01% μπορεί να φαίνεται τεράστιο άλμα για τους αλείς. Δεν έχουν όμως έτσι τα πράγματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες περισσότερες περιοχές όπου δεν υπάρχουν ελευθερικές δραστηριότητες. Ίσως να κάνουμε κάποιο λάθος, αλλά ε, αυτό εδώ το θέμα της, ε, της, της ε, χωροταξίας της θάλασσας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Σάτων έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση γιατί αισθάνθηκα κάποια σύγχυση. Νομίζω ότι διάβασα στην πρώτη διαφάνεια ότι η περιοχή των χωρικών διδάτων περιορίζεται στα 12 μίλια. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές, αυτές τις υποχρεωτικές ε, ε, ζώνες προστασίας μέχρι 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια από την ακτή. Σίγουρα δεν το είδα αυτό σε καμία τροπολογία που κατέθεσαν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα τις ψηφίσουμε εν το χρόνο. Αλλά είχα κάποια δυσκολία διότι νομίζω ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια όσον αφορά την ε, προσέγγιση του κειμένου σχέση με κάποιες από αυτές τις τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι μιλάμε για 8 έως 12 μίλια. Ή νόμιζα ότι έτσι ισχύει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια έρευνα όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτού του μέτρου σε περιοχές όπως είναι η Σκοτία. Ποιος θα είναι ο οικονομικός ε, ε, αντίκτυπος στην, ε, θα είναι στη Δυτική Σκοτία από 0 έως 12 μίλια αν εφαρμοστεί και αν θα είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή. Και θα είναι, ε, δεν θα υπάρξει θα είναι δυσανάλογος αν την εφαρμογή της Σκοτίας σε σχέση με άλλες περιοχές της Αγγλίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι εκ των υστέρων για να σταθμίσουμε αυτούς τους αντικτύπους. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν αρκετά κονδύλια στον Ταμείο Αλίας, εφόσον υπάρχει υποχρεωτική εφαρμογή σε ορισμένες περιοχές. Γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εδώ αυτό το οποίο θα συμβεί είναι αν εφαρμοστεί αυτό ε, θα ισχύσει για πάντα. Οι τροπολογίε λένε ότι θα πρέπει να ισχύσει για πέντε χρόνια, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να κλείσει μια άλλη περιοχή για άλλα πέντε χρόνια. Άρα μιλάμε για μια εφαρμογή στο διενικέ. Και τελικά δεν θα είναι δυνατόν ε, να αντέξουμε το οικονομικό κόστος. Και θα είναι εις βάρος των αλλίων. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και δεν νομίζω ότι ακούσαμε εδώ αρκετά πράγματα, ούτε ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προφανή ωφέλη της διατήρησης των αστακών και τον αντίκτυπο που θα έχει σε κάποια είδη τα οποία είναι υψηλή κινητικότητας. Όταν μιλάμε για τα από 0 έως 12 μίλια υπάρχει και ένα άλλο θέμα Ε, το οποίο αναφέρεται σε ορισμένε από τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ορισμένες χώρες μέλη θα πρέπει και οι περισσότερες ε, συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής αφορούν την αποκέντρωση. Ενώ εδώ υπάρχει μια αντίθετη τάση υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κεντρωτικού, κεντρικού μέτρου. Ε, παράλληλα έχουμε αύριο μια ψηφοφορία εν σχέση με την ε, διεύρυνση αυτού του καθεστώτος. Θα εφαρμοστεί αυτό λοιπόν στο όριο των 12 μιλίων σε άλλες περιοχές εκεί που τα πράγματα λειτουργούν ε, καλά. Ενώ υπάρχουν ε, άλλα θέματα όπου η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις περιοχές. Εμένα δεν ε, με καταπλήσουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αλλά θεωρώ ότι δεν, έχουν, δεν παρέχουν καμία απάντηση οι τροπολογίες εν σχέση με το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την ε, ζώνη των 12 μιλίων. Για παράδειγμα, όσον αφορά το μέτρο των ε, συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσει. Και όσον αφορά ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο αναφέρθηκε από ορισμένου ε, βουλευτέ ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε ορισμένε περιοχέ, σε ορισμένε κοινότητε. Και μια από τι δυσκολίε είναι το πώς θα την ερμηνεύσουν οι αλληλείς. Για παράδειγμα, είπαν ορισμένοι βουλευτέ ότι δεν θα υπάρχει καθόλου αλληλευτική δραστηριότητα στην περίπτωση αυτή τη περιοχή αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πείσει ωστόσο τους σε αυτές τις περιοχές θετικής σκοτίας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καθόλου αλληλευτική δραστηριότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πιστούν. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πάμε σε αυτούς τους, ε, στους αλείς και να τους ε, πούμε ότι υπερψηφίσαμε αυτά τα μέτρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε τις αλευτικές μας κοινότητες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ, είναι η διατύπωση των τροπολογιών και ο υποχρεωτικό ε, χαρακτήρα αυτή τη συγκεντρωτική πολιτική, ενώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία αποκέντρωση σε σχέση με αυτέ τι αποφάσει. Thank you κυρία Λέβιν, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ρόμπερτς, για την εξαιρετική έκδοσή σας και την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική, γιατί είδαμε παραδείγματα ανά των κόσμων για το τι μπορεί να κάνουμε με τα αποθέματα των στις προστατευόμενες περιοχές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα είδη τα οποία είναι σε μετακίνηση μπορούν να είναι εκτός προστατευόμενης αίριας, αλλά και εντός των προστατευόμενων περιδών έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, να, αφού υπάρχουν λοιπόν και εντός και εκτός πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος και για τα αλλιεύματα λέει και για τους ίδιους τους αλείς. Μιλήσατε για ένα δέκατο της χιλής στη Μεσόγειο. Πολύ μικρό ποσοστό. Το ίδιο συμβαίνει και τη χώρα μου, την Σουηδία, όπου έχουμε πάρα πολύ λίγες μικρές αλληλευτικές περιοχές, στις οποίες δεν αναπτύσσονται αλληλευτικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους στόχους της Ναγκόγια. Πριν από δύο χρόνια στην Ναγκόγια, στην ε, Ιαπωνία, ο κόσμος απεφάσισε και προσυπέραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 10% των ε, αλλιευτικών πόρων να το προστατεύσουμε. 10% λοιπόν για τα θαλάσσια, πιστεύουμε ότι είναι 10%. Αλλά αν το συγκρίνουμε με τα είδη τα χερσαία, όπου έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, δεν είναι μεγάλο. Είδαμε σε 200 χρόνια πώς άλλαξαν τα πράγματα και είδαμε πόσο πρέπει να προστατεύουμε τη χλωρίδα και την ε, πανίδα. Είναι λοιπόν φυσικό να θέτουμε τέτοιου είδους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Δεν πιστεύω, αλλά ο κύριος Μιλάνα, αν κάνω λάθος θα με διορθώσει. Δεν νομίζω ότι η τροπολογία του κυρίου ε, Μιλάνα είχε στόχο μόνο τα 12 ναυτικά μίλια στις προστατευόμενες, στις προστατευόμενες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας να υλοποιήσουμε τους... αυτά τα οποία λέγονται στη Συμφωνία της Ναγκόγια και να τα αποθ... αλλιευτικά μας αποθέματα. Μία ερώτηση στον κύριο Ρόμπερτς. Πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί δίκτυο μεταξύ αυτών των προστατευόμενων θαλασσίων περιοχών, διότι με αυτή τη δικτύωση θα ξέρουμε πώς ακριβώς τα πράγματα. Αν έχουμε μία ζώνη εδώ και μία άλλη αλλού, ίσως δεν επιτυγχάνονται πολλά πράγματα. Πόσο σημαντική είναι λοιπόν Όπω Όπως είπε και ο κύριος Μιλάναμ, η προστασία αυτών των ε, ζωνών όπου έχουμε τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση αλίας είναι κάτι το οποίο γίνεται και θα βοηθήσει και τελικά, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το να έχουμε μερικώς προστατευόμενες περιοχές γύρω από τις αμυγός προστατευόμενες ε, περιοχές είναι εξαιρετική ιδέα. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία πάντα προσπιζόμαστε ως αρχή στην Επιτροπή μας. Δηλαδή, ότι γίνει να γίνεται και προς όφελος τις της αλληλευτική ε, βιομηχανίας και των αλλήλων. Ο κύριος Τόβαλτ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε τον κύριο Τόβαλτ την εκθεσή του. Λέμε στα γερμανικά γιατί να το κάνουμε απλά όταν μπορούμε να το κάνουμε πολύ σύνθετα. a little for you. Θα σας πω λοιπόν και εγώ κάτι απλό πολύπλοκο, επειδή κανένας δεν σας το είπε μέχρι τώρα με αυτό που λέω. Υπάρχουν ε, οι οικολογικές διαδικασίες που δεν ελέγχονται, άλλες που ελέγχονται. Και ως παράδειγμα θα πω το εξής μείωση του ποσοστού άλατος στην Βαλτική. Σχέση με το τι γίνονταν από 30 χρόνια. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, είναι εκτός θέματος αυτό. Αυτή η μείωση λοιπόν της αλατότητας, του ποσοστού του άλατος. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει όλη την διαδικασία, το είδος του αλλιεύματος. Υπάρχουν προβλήματα με τον ε, γάδα, με τον μπακαλιάρο, εξαιτίας αυτής της αλλαγής του ποσοστού άλατος, της αλατότητος, uh, για πολλούς λόγους. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς μπορεί κανείς να αποκαταστήσει αυτή τη ζώνη αλλή όταν πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή την κατάσταση και όταν υπάρχουν όλες αυτές οι αλλαγές. Στη Βαλτική, λοιπόν, πώς μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αποκατάσταση όταν τα αλλιευόμενα ήδη αλλάζουν εξαιτία αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Επιτροπή. Uh, just to say, I mean, the, Commission welcomes the report. Ήθελα απλά να πω ότι η Κομισιόν υποστηρίζει και την έκθεση και τις συστάσεις. Απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να τη μελετήσουμε. Ένα σχόλιο μόνο. Ενώ υποστηρίζουμε την ιδέα αυτών των προστατευόμενων περιοχών μεγάλου μεγεθού, πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει αυτό να συμπληρωθεί με μια ισχυρή πολιτική σε θέματα ικανότητα, χωρητικότητα, ε, ώστε αυτέ οι προστατευόμενες ε, περιοχές να μην γίνουν ε, περιοχές όπου θα πηγαίνουν όλα τα σκάφη και θα ψαρεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε με υποστήριξη της ελευτικής προσπάθειας και για να μην έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Ρόμπερτ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, στις απαντήσεις που θα δώσω σε όλες αυτές τις εξαιρετικές ερωτήσεις και τα σχόλια που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τα κόστη. Σίγουρα η δημιουργία τέτοιων περιοχών, οποιοδήποτε είδους, ε, κοστίζει πολλά. Χρειάζεται διαβουλεύσεις, συμμετοχή των κοινοτήτων, ε, ερευνητικό έργο και ούτω καθεξής. Αυτές ωστόσο οι δαπάνες ε, θα μας επιστραφούν πίσω με τα ωφέλη που θα παράγουν αυτές τις περιοχές. Ε, ε, μια μελέτη μεσογειακών προστατευόμενων περιοχών που εξετάζει τα ωφέλη για τον τουρισμό και την αλληλεία, το τομέας του τουρισμού εννοώντας τις καταδύσεις, τις ψυχαγωγικές καταδύσεις και την ψυχαγωγική αλληλεία. Τα ωφέλη λοιπόν από αυτές τις προστατευόμενες περιοχές ε, ήταν ε, το διπλέ, διπλές από το κόστος δημιουργίας αυτών των προστατευόμενων περιοχών. Είναι λοιπόν ένα διαχειρισμό κόστο και αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Μπορούμε να αναμένουμε ότι η δαπάνη θα μειώνεται με το χρόνο σε σχέση με την, καθώς θα αυξάνονται τα ωφέλη. Ρωτήσατε πώς αγοράζει κανείς ε, την υποστήριξη της αλληλευτικής βιομηχανίας. Πολύ λοιπόν μίλησαν για τι δαπάνε τη αληθική βιομηχανία, για το κόστο αυτό τη αληθική βιομηχανία, Ο τρόπο με τον οποίο αγοράζει κανεί την υποστήριξή του, είναι βοηθώντα του κατά τη μεταβατική περίοδο. Τι συμβαίνει όταν δημιουργούμε μια προστατευόμενη περιοχή, εντό ενό ενός-δύο ετών τα πράγματα δυσχεραίνουν για όσου εργάζονται στην αληθική βιομηχανία προσπαθώντα να βρουν νέε αληθικέ περιοχέ καθώς ε, τα ωφέλη ε, από την αποκατάσταση των ηχθείων αποθεμάτων ακόμη βρίσκονται υποδημιουργία. Χρειάζεται Χρειάζονται λοιπόν υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον. Ε, ενώ υφίστανται τα το βραχυπρόθεσμο κόστος της δημιουργίας αυτών των περιοχών. Στο σώνοφορο αφορά το σχολείο του κ. για αυτές τις δαπάνες που θα συνεχίσουν επάπειρον, δεν θα συνεχίσουν επάπειρον Ειδικότερα αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ότι οι δαπάνες, το κόστος θα μειώνονται με το χρόνο καθώς θα αρχίσουν να συσσωρεύονται τα ωφέλη. Έτσι λοιπόν οι ευκαιρίες αλληλείας θα, θα αυξηθούν σταδιακά γύρω από αυτές τις περιοχές ε, προστασίας ε, αποκατάστασης εχθεία αποθεμάτων. Όπως είπα λοιπόν είναι μια επένδυση στο μέλλον των ανθρώπων παρά κάτι που θα τους αφαιρεί κάθε έτος ε, πόρους. Ουσιαστικά δημιουργούμε μια επένδυση η οποία θα αναπτύσσεται με τον χρόνο ακριβώς όπως και οποιαδήποτε άλλη οικονομική επένδυση. Όσον αφορά τα ποσοστά, τα ποσοστά είναι λίγο ασαφή στην πρόταση. Αυτά τα ποσοστά θεωρείται ότι πρέπει να είναι 10 20%. Τι ξέρουμε τώρα. αν πρέπει να στοχεύουμε το 20% 30% το οποίο επίσης δικαιολογείται από όλα τα επιστημονικά στοιχεία που κυκλοφορούν, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι το 1-2% που κάνει τη διαφορά και σίγουρα δεν είναι το ένα χιλιοστό της θάλασσας που πρέπει να προστατεύουμε από την εκμετάλλευση. Αν θέλουμε σημαντικά ωφέλη για την ελληνική βιομηχανία πρέπει να περάσουμε από αυτές τις μικρές προστατευόμενες περιοχές που μελετούσαμε μέχρι σήμερα και να φέρουμε αυτές τις περιοχές τουλάχιστον στο 10% των θαλασσιών περιοχών. Και ποιο ρώτησε τι γίνεται στις μικρές χώρες που συμβάλλουν με μεγάλο κομμάτι της οικονομικής τους δραστηριότητας και πώς θα υλοποιηθούν τα πράγματα αυτά σε όλα τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω εγώ ότι είναι ισότιμα, έχει νόημα όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην επιτευξή αυτής της πολιτικής. Αλλά κανένα κράτος μέλος ε, δεν θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ή σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα, διότι το 20% του Βελγίου είναι το ίδιο με το 20% της Σκοτίας ή το 20% της Δανίας η συνολική περιοχή είναι μεγαλύτερη, αλλά το κλάσμα που αφιερώνει κανείς σε αυτά τα μέτρα ιδιαίτερη είναι το ίδιο, το ποσοστό. Το θέμα είναι ότι εάν ε, οι χώρε δεν καθιερώσουν αυτέ τι περιοχέ, αυτό που γνωρίζουμε ότι θα γίνει δεν θα αποκομίσουν τα ωφέλη, τα τοπικά ωφέλη αυτών των προστατευόμενων περιοχών. Και όπω είδαμε, τα ωφέλη αυτά παρέχονται τοπικά, όπω ε, διαπιστώσαμε σε προστατευόμενε περιοχέ στην Ισπανία και σε άλλε περιοχέ. Ακούσαμε μια διευκρίνηση για το ποσοστό αύξησης ε, των αλλιευμάτων στις γύρω περιοχές κατά 2 με 4%. 2,4% έτος με έτος. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι αυτό το όφελος αυξάνεται με το χρόνο. Δεν είναι ότι κάθε χρόνο έχεις όφελος 2-4% και αυτό είναι όλο ή ε, μάλλον τον πρώτο χρόνο έχει 2,4% και αυτό είναι όλο. Αυτό το όφελο αυξάνεται με το χρόνο ω αποτέλεσμα αυτή τη βαθμία συσσόρευση ε, ε, αυξήσεων 2 με 4% των ελευμάτων κάθε χρόνο. Και το άλλο που έχω να πω είναι ότι όταν συγκρίνει κανεί τα ωφέλη αυτών των προστατευόμενων περιοχών, πρέπει να εξετάσουμε τι συμβαίνει σε περιοχέ μη προστατευμένε. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει δυστυχώ πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι τα αλλιεύματα βρίσκονται σε ευθύνουσα πορεία. Ε, αν προστατεύσουμε λοιπόν αυτές τις περιοχές και δημιουργήσουμε ωφέλη, η διαφορά μέτρησης είναι μεταξύ ουσιαστικά του status quo, της, της αυτής, αυτό το φθήνο status quo και αυτή την αύξηση. Αυτά τα δύο συγκρίνουμε. Δηλαδή το όφελος ε, ενδεχομένω ακόμη μεγαλύτερο αν το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Επίση τέθηκε το ερώτημα των μερικώς προστατευόμενων περιοχών, πόσο μεγάλες πρέπει να είναι. Αυτέ οι μερικώς προστατευόμενες περιοχές μπορούν να είναι όσο θέλουμε. Συνήθως όμως πρόκειται για περιοχές ε, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση σκάφη με εξοπλισμό που δημιουργεί μεγάλη ζημιά. Μιλάμε τώρα για κινητού εξοπλισμού όπω στρατεσβηθού, γάρι δαλευτικά που δημιουργούν που προκαλούν τα χειρότερα τις χειρότερες συνέπειες ε, αυτές οι περιοχές λοιπόν προστατεύονται από αυτά τα είδη εξοπλισμού τώρα το κατά πόσο θα πρέπει να συμμετέχει ο τομέας ε, των αλλιέων ε, η βιομηχανία, η ελευτική βιομηχανία ναι συμφωνώ πρέπει να συμμετέχει τα μειονεκτήματα της συμμετοχής ή ε, της ανάθεσης της απόφασης στην ελευτική βιομηχανία είναι ότι η της αναθεσης της αποφασης στην αλληλευτικη βιομηχανια ειναι οτι η ελαχιστοποιηση του κόστους βραχυπρόθεσμα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση αυτών των περιοχών όσον αφορά την απόδοση, την αποκατάσταση των ελευμάτων. Χρειάζεται λοιπόν μια ισόρροπη διαδικασία μεταξύ ελεκτικής βιομηχανίας και επιστημόνων για να μπορέσουν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Το ερώτημα του πώς σε επενδύσεις χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλα αυτά δεν είναι αμεληταίο ποσό. Αλλά δεν είναι και δυσανάλογο. Ε, αν το δούμε σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που πληρώνουμε για την αλληλεία, ε, είναι μάλλον μια ικανοποιητική επένδυση, μάλλον θα έλεγα ευκαιρία όσον αφορά αυτά τα κόστη. Για σας δώσω το παράδειγμα της Καλιφόρνιας, όπου σε ολόκληρη την πολιτεία υπάρχει ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που καλύπτει 16% των ε, υδάτων της Καλιφόρνια. Αυτό κόστησε 37 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών. Σημαντική λοιπόν επένδυση, αλλά έχουν τώρα ενός ύψους του επίπεδου δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που εγώ θεωρώ πιο συναρπαστικό για... εκπονώντας αυτή την έκθεση εξετάζοντας τη πιο πρόσφατη βιβλιογραφία για τις περιοχές αποκατάστασης ηχθεία αποθεμάτων και βρίσκοντας ε, πώς λειτουργούν τα αποτελέσματα που παράγουν, ποια είναι τα ωφέλη για την ελληνική μηχανία ποια είναι το κόστος για την ελληνική βιομηχανία, διότι την τελευταία φορά που είχα κοιτάξει τα στοιχεία ήταν το 2002. Τότε δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο λεπτομερή. Είναι αρκετά για να αποτελέσουν μια σταθερή βάση για χάραξη πολιτική εδώ. Ο κ. Μιλάνα μίλησε για πληρωμή προς ανθρώπους ώστε να μην ψαρεύουν. Αυτό το βλέπουμε συχνά στη Γεωργία, όπου καταβάλουμε χρήματα σε κάποιους για να μην χρησιμοποιούν εδάφη είναι μια προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστου δημιουργία προστατευόμενων περιοχών ε, σε διάφορε περιοχές και στη θάλασσα, όπως το Great Barrier Reef, όπου υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η, η, εκεί έλαβε αποζημίωση για την απώλεια ε, αλληλευτικών περιοχών. Ε, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν... Ε, ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Αλίας και Θάλασσας ε, για τέτοιες αποζημιώσεις. Αυτό ανταπαντά και στο σχόλιο της Επιτροπής ότι δεν είναι η λύση των, όλων των προβλημάτων αλίας στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της λύσης. Αποτελεί ένα σημαντικό θεμέλιο για οτιδήποτε άλλο καλό θέλουμε να κάνουμε στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, τη μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας, τα μειωμένα απόβλητα λόγω απορρίψεων ε, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι προτάσεις που ε, πρέπει επίσης να εφαρμοστούν ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική αλληλευτική πολιτική στην Ευρώπη. Προερχόμενος τώρα στον κύριο Χάτο, μιλήσατε για τις επιπτώσεις μια πολιτική τέτοιου είδου, για μικρές κοινότητες που εξαρτώνται από την Αλία στη Δυτική Σκοτία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι κοινότητες υποφέρουν από την υπεραλίευση. Έχω μελετήσει τις επιπτώσεις της υπεραλίευσης στη Δυτική Σκοτία λεπτομερώς. Έχουν χάσει πάρα πολλά αυτές οι κοινότητες ε, που βασίζονται στην αλληλεία και πλέον έχουν ελάχιστα πράγματα να λεύσουν, μόλις κάτι τρακόδραμα. Και αυτό που χρειάζονται είναι σημαντική προστασία από τους κινητούς εξοπλισμούς ε, που χρησιμοποιούνται. Ε, τα πρώτα βήματα που χρειάζονται για την αποκατάσταση αυτών των κοινοτήτων είναι η υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Αυτή η αποκατάσταση θα είναι σταδιακή, οι αλληλευτικές ευκαιρίες ε, θα βελτιωθούν με το χρόνο και αυτό θα επιλύσει κάποιες έχεις μεταξύ διαφορών αλληλευτικών τομέων που παρατηρούνται στην αλληλεία της Ευρώπης και που αυξάνονται, με το χρόνο λόγω των διαφόρων προβλημάτων. Αυτό θα βοηθήσει λοιπόν ε, στον έλεγχο των κινητών και σταθερών εξοπλισμών στην Αλία. Μιλήσαμε για το στόχο της Ναγκόια. Είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αλία έχει επηρεάσει τα είδη και τους οικότοπους στα ευρωπαϊκά ύδατα σε τεράστιο βαθμό και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να επαναφέρουμε την αρχαίγονη κατάσταση των ευρωπαϊκών θάλασσεων πρέπει να κοιτάξουμε πριν 300 χρόνια πριν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει την εξάλληψη πολλών ειδών από μεγάλες θαλασσίες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Μεγάλα, πολλά ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Ήταν ε, ψάρια που υποστήριζαν παραγωγική αλληλεία όπως ο Καρχαριάς Άγγελος και ε, Κάποια από αυτά τα είδη έχουν ήδη εξαφανιστεί, είναι υπό εξαφάνιση. Η εφαρμογή λοιπόν τέτοιων τοποθεσιών αποκατάστασης εκθεαποθεματων είναι ένα σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων εξαφάνιση ορισμένων ειδών και ταυτόχρονα των ποσοτήτων. Τώρα η επίτευξη των μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων μέσω αυτών των περιοχών πιστεύω θα επιταχυνθεί η αποκατάσταση θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Ο ταχύτερο τρόπο επίτευξη του MSB είναι να σταματήσουμε να ψαρεύουμε οπουδήποτε, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο επόμενο καλύτερο τρόπο είναι η δημιουργία περιοχών προστατευόμενων από οποιαδήποτε αλεία και η διατήρηση των υπολείπων περιοχών ανοιχτών στην αλία και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονα ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις Μόνο βραχή πρόθεσμα για την ελληνική βιομηχανία μίλησαμε. Μίλησε ο κ. Τόρβαλτ για τις τεράστιες οικολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Ε, δεν το έχουμε πει, αλλά ένα από του σημαντικότερου λόγου για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, παρέχοντα περισσότερη προστασία στι ευρωπαϊκέ θάλασσε και αυξάνοντας την ποιότητα των θαλασσών είναι να έχουμε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέχρι το 2020, αλλά οι θάλασσες σήμερα βρίσκονται υπό σημαντική πίεση όχι μόνο λόγω της αλίας, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ρήπανσης, της ε, ε οξύδους των ωκεανών. Ε, έχουν, υφίστανται τεράστια πίεση με, με πολλούς τρόπους. Ε, Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αλίας, βοηθάμε τη θάλασσα να γίνει πιο... Ε, να έχει μεγαλύτερη αντοχή. Δίνουμε στο θαλάσσιο περιβάλλον μια δυνατότητα να προσαρμοστεί και να καταπολεμήσει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η οξύτητα των υδάτων, για παράδειγμα. Πρέπει να ανεβάσουμε λίγο λοιπόν, λοιπόν την παρά, πρέπει να αυξήσουμε την αυθονία των ψαριών στη θάλασσα, το ποσοστό πολλαπλασιασμού αυτών των αποθεμάτων, ώστε να αποκτήσουν ε, την αντοχή που χρειάζονται όλα αυτά τα είδη, ώστε να αντιμετωπίσουν τι αλλαγέ, διότι τα πράγματα πρόκειται να επιδεινωθούν αρχικά και μετά θα βελτιωθούν. Θα χρειαστούμε χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω τη αύξηση του ανθρωπινού πληθυσμού, και τη κλιματική αλλαγή και όλων των ζητημάτων που προκαλεί. Πού θα βάλουμε αυτές τώρα τις προστατευόμενες περιοχές. Το ευκολότερο που μπορούμε να σκεφτούμε βάσει μιας επενδυτικής στρατηγικής, όπως σε κάθε επενδυτική στρατηγική που δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον καθαρά, τι θα έκανε ένας επενδυτής τραπεζίτης που θα βαλουμε αυτέ τωρα τις προστατευομενες περιοχέ. το ευκολοτερο που μπορουμε να εξαπλώσει, μια επενδυτική διαδώσει τους κινδύνους, ε, την επικοινωνία. Δεν επενδύει ένα επενδυτή τραπεζιτη που θα προσπαθησει να εξαπλωσει να διαδωσει του κινδυνους την επικοινωνια δεν επενδυει κανεί ολα τα χρήματα σε ένα είδος ομολόγων. Ε, επενδύει τα πράγματα σε διάφορα σε διάφορους τίτλους ώστε να έχει περιορισμένο κίνδυνο. Τι γίνεται λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με τι προστατευόμενε περιοχέ. Τι δημιουργούμε σε διάφορα μέρη, δεν τι βάζουμε όλε στο ίδιο μέρο, ελπίζοντα ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Τι εξαπλώνουμε σε, στα ευρωπαϊκά ύδατα, σε πολλέ διαφορετικέ περιοχέ και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι ω δίκτυο θα έχουν καλή απόδοση μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ο πλούστερο τρόπο για να το εξετάσει κανεί. Όσον αφορά τώρα τα δίκτυα, όπως στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Λαβρή, είναι σημαντικό να έχουμε αυτέ τι προστατευόμενε περιοχέ ω δίκτυο, από τη μορφή δικτύου, διότι ανά πάσα δεδομένη στιγμή Ορισμένε περιοχέ δεν θα έχουν τόσο καλέ αποδόσει όσο άλλε και αυτέ υποστηρίζονται αμοιβαία μεταξύ του ε, εφόσον υπάρχει τέτοια ανταλλαγή αυγών και προνυμφών. Ε, Εάν λάβει κανείς υπόψη αυτά τα μοτίβα αλληλοσύνδεσης, αυτό που, που μπορούμε να προτείνουμε είναι να, να έχουν διαστάσεις 10 με 12 χιλιόμετρα, σε να έχουν μέγεθος 10-12 χιλιόμετρα σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων διάφορα επιστημονικά συμπεράσματα μας οδηγούν σε αυτό τον εμπειρικό κανόνο. Αν έχουμε ε, καταφύγια μεγέθους 10 χιλιόμετρων σε αποστάση 80 χιλιόμετρων, έχουμε το χαμηλότερο, το χαμηλότερο κινδύνο. Ουσιαστικά έχουμε διάφορα, διάφορα εύρη ε, μεγέθους τέτοιων προστατευόμενων βρεχών και απόσταση μεταξύ τους που μπορούμε από το λιγότερο επικίνδυνο μέχρι το πιο επικίνδυνο. Θα μα βοηθήσουν να αυξήσουμε τη ζωτικότητα και την αντοχή και ε, την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Μου ζήτησαν ε, το λόγο δύο συνάδελφοι, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κύριος Αρσένης. Ναι, καταρχήν, σε σχέση με τα όσα είπε ο εισηγητής, αφορά την ε, παράκτια περιοχή, μόνο τα 12 μίλια. Και επίσης, η ιδέα αυτή ως έχει περιλαμβάνει όλες τις άλλες περιοχές που είναι κλειστές. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν αυτά τα αεολικά πάρκα. Παρόλο που εκεί ε, μπορεί ε, να είναι, ε, το έδαφος μπορεί να είναι, να είναι τέλματα ή να μην ενδείκνυται για να μην είναι ιδιαίτερα εύφορα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική παρατήρηση για την ε, Δυτική Σκοτία. Ο μιλητής ε, είπε ότι μεγάλο τμήμα της, ε, των αλλιέων εξαρτώνται από αλεύματα υψηλής αξίας και από γαρίδες και χένια. Ε, τώρα, όσον αφορά το κόστος αυτής της ε, πρότασης, θεωρώ ότι το κόστος θα είναι δυσανάλογο εάν ε, εφαρμοστεί στην περιοχή αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία και εν σχέση με το εκτιμόμενο κόστος για μια περίοδο πέντε ετών. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάτον. Ο κύριος ε, Μιλάνα έχει το λόγο. Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι πρωτοβουλία για την διατήρηση, αλλά... Αλλά το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε τους πόρους. Ίσως πρέπει να το, να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά δεν είναι μόνο το θέμα να ε, συντηρήσουμε αλλά και να διαχειριστούμε τη θάλασσα. Είναι άλλη έννοια. Δεύτερον, ε, πρέπει να υπάρχει ομοιογενής ε, κατανομή, διότι αν δεν είναι ομοιογενής θα δημιουργήσει πλούσιους και φτωχούς. Αυτή η ομοιογένεια και η συνεργασία, αν δεν υπάρχουν, καταλύουν οποιαδήποτε δομή. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μέτρο συντήρησης των δραστηριοτήτων μας, αλλά διαχείρισης. Ο κύριος Ρόμπερτς. Yes, uh, so, so very brief. Ναι. Θα είμαι σύντομος. Ε, ξέχασα να αναφερθώ στις de facto προστατευόμενες περιοχές και ποια θα μπορούσε να είναι η δική του συμβολή στο συνολικό δίκτυο των περιοχών αποκατάστασης των ηχθιακών αποθεμάτων. Αναφερθήκατε στα ελληνικά πάρκα. Σε σχέση ε, με τα κινητά αληφτικά μέσα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ε, ε, αναβάθμιση των αλευτικών περιοχών. Ε, πράγματι οι περιοχές αυτές ε, είναι περιοχές αποκατάστασης των ελευτικών αποθεμάτων. Είδαμε ποια είναι τα αποτελέσματα ε, στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά το θέμα του οικονομικού προϋπολογισμού, όσον αφορά το θέμα αυτό που αναφέρατε για τα χτένια και τις ε, γαρίδες και τα ποσοστά αυτά. Η δική τους ε, ε, σημασία είναι φθήνουσα. Και αν δούμε την αύξηση αυτής της βιομηχανίας οστρακόδερμων και τη φθήνουσα τάση από την άλλη, ορισμένων τύπων αλίας, ορισμένων αλιευμάτων, συγγνώμη. Με τον τρόπο αυτό μετακινούνται τα νεογνοί και αλλάζουν τους ε, οικοτόπους. Έτσι λοιπόν ε, τα... Ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές τις περιοχές από τα ψάρια. Για να έχετε λοιπόν μια αποκατάσταση των νυχτιακών αποθεμάτων θα πρέπει να τεθούν κάποια όρια σε αυτούς τους ε, πληθυσμούς ε, από γαρίδες και χτένια. Έγινε μια έρευνα στη Δυτική Σκοτία η οποία δείχνει ότι η αποκατάσταση της ε, ποικιλία αυτών των ψαριών θα αύξανε τη συνολική αξία της αλίας σε όλη τη Δυτική Σκοτία ως αποτέλεσμα αύξησης στον ε, τομέα αλίας που γίνεται με σταθερά αλληλευτικά μέσα, αλλά και την αναζωγόνηση των αποθεμάτων. Γιατί είχαμε απόλυτα τα πρωτογενή αποθέματα μέχρι 60 τόνοι ψάρια εκφορτώνονταν και ε, πριν από λίγο καιρό τελικά, ε, πριν από μερικά χρόνια εξαφανίστηκαν εντελώς τα αποθέματα των νυχθείων. Δεν υπήρχαν πια ψάρια να ληφθούν. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να διευρυνθεί η οικονομική βάση αυτών των περιοχών, όπως είναι η Δυτική Σκοτία, αντί να παραμένει εξαρτημένη από ορισμένα είδη αλίας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτού του θέματος και περνούμε στο επόμενο. το οποίο είναι ειδική ορή όσον αφορά την αλληλεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό και διατάξεων αφορά την αλληλεία σε εθνή υδά του Βορειοδυτικού Ατλαντικού και κατάρριση του κανονισμου αριθμό αριθμός 2347-2002. Η συγκητή έκθεση αυτή είναι ο κύριο Ασένης. Σήμερα θα κάνουμε την παρουσίαση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματο αυτού Γι' αυτό δίδω αμέσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φρίς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα παρουσιάσω την πρόταση της Επιτροπής. Ο κανονισμός έχει ως στόχο με να αλλιεύουμε τα αποθέματα βαθέων υδάτων με τρόπο βιώσιμο, ώστε τα υπεραλλιεύματα και τα by catches, οι απορρίψεις, να μην είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί πρόβλημα στην ισορροπία. Παρακαλώ, ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί προτείνουμε κανονισμό για τα αποθέματα βαθέων υδάτων, διότι πρόκειται για μια ειδική αλία. Μιλούμε για βάθος από 600 έως 2 με 3.000 μέτρα και μέχρι τώρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για το πότε και πώς αλλιεύουμε σε αυτές τις περιοχές και αντιμετωπίζουμε συχνά μια κατάσταση στην οποία δεν κατανοούμε ούτε εμείς ούτε πλήρως οι επιστήμονες. Ξέρουμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες γνώσεις. Επίσης τα αποθέματα βαθέων υδάτων είναι πάρα πολύ ευάλωτα διότι αναπαράγονται και αναπτύσσονται πάρα πολύ αργά. Φτάνουν την οριμότητα αργά στη ζωή τους και εάν τα αλλιεύσουμε πολύ νέα και αν δεν κάνουμε αλληλεία ε, αηφόρο, τα αφανίζουμε. Τα οικοσυστήματα λοιπόν, επίσης, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Έχουμε κοράλια, έχουμε σφουγγάρια. τα οποία μπορεί από την αλία να καταστραφούν Αυτή όμως του είδου η αλληλεία είναι μια δραστηριότητα, τίποτε δεν μπορούμε, δεν μπορούμε ότι 100% πρόκειται για κάτι λανθασμένο. Υπάρχουν οι κανονισμοί, υπάρχουν οι ποσοστώσεις, όπω και σε άλλου τομείς. Έχουμε τέτοιου είδου ε, βαθύβια αλλιεύματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, όπως φυρίδες, συναγρίδε ή δεν ξέρω τι άλλα παρεμφερεί. Αλλά πρέπει ότι κάνουμε ως δραστηριότητα να το κάνουμε με αηφόρο τρόπο. Δεν θέλουμε με την πρότασή μας να απαγορεύσουμε, ούτε να περιορίσουμε την αλία βαθέων υδάτων, αλλά να βρούμε τρόπους που θα την κάνουν διαχειρίσιμη όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και των αποθεμάτων. Ο στόχος μας είναι, εδώ είπαμε, τα λιεύματα βαθέων υδάτων. Στον κανονισμό υπάρχουν οι ορισμοί για να ξέρουμε με τι είδους, ε, τι είδους αλλιεύματα καθορίζουμε, τι είδους αλλιευτικά σκάφη, σε τι είδους αλλιευτικά σκάφη αναφερόμεθα και επίσης καθορίζονται ε, τα είδη εργαλείων και δικτυών τα οποία χρησιμοποιούνται απλά για τα δίχτυα βυθού για να μην γίνονται καταστροφές και πώς σιγά σιγά μπορούμε τις στράτες ε, αυτές τις βαθίες αλίας σιγά σιγά να τις αντικαταστήσουμε για να μην καταστρέφουν τα αλλιεύματα. Επίσης υπάρχει πρόταση για τη βελτίωση του πλαισίου για την συλλογή δεδομένων που αφορούν αυτή την αλία βαθαίων υδάτων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πρότασης αυτής οικονομικής πλευράς και για την αλλιευτική βιομηχανία. Οι επιπτώσεις των ε, βορειοανατολικό Ατλαντικών είναι περιορισμένος. Έχουμε ποσοστό 1% των αλλιευμάτων μόνον, που είναι τέτοιου είδους αλλιεύματα από ε, βαθέων υδάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όσον αφορά τα ανώτατα ε, επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ως παράδειγμα, αν δείτε όμως άλλες περιοχές, όπως το Λοριόν στη Γαλλία, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια αλλιευτικά σκάφη που κάνουν αυτού του ίδιου ε, είδους την αλλιεία. που αναπτύσσουν και άλλες ε, δραστηριότητα, αλλά εφόσον χρησιμοποιούν εξοπλισμό και τεχνικές μικτές, γιατί κάνουν και άλλους αδεία, πρέπει να την ε, τροποποιήσουν, να την προσαρμόσουν. Με ποια μέσα, με το μέσο που προβλέπουμε εμείς για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να γίνουν αλλαγές στον εξοπλισμό, στα λιευτικά σκάφη και όλα αυτά στα πλαίσια του νέου MMF. Πριν να ολοκληρώσω, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Γίνονται συζητήσεις και αυτό και με τους επαγγελματίες του κλάδου και με τους αλλοίς το ακούμε ότι εκφράζονται φόβοι και πιστεύουν κάποιοι ότι μια τέτοια πρόταση έτσι όπως έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή ίσως είναι το πρώτο βήμα προς την ε, απαγόρευση τέτοιου είδους στρατών ε, βαθύβιας Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ήδη αναφέρεται σε αγωγικές παρατηρήσεις. Η πρόθεση της πρότασης δεν είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Και το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά αυτή την αλία βαθέων υδάτων αναφέρεται σε ειδικέ περιπτώσεις συγκεκριμένε, και δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα ή προβλέψεις για άδου ε, είδους ε, ε αλληλεία που χρησιμοποιεί τράτες βυθού. Αναφερόμαστε μόνο στην αλληλεία βαθέων υδάτων. Αυτά ήθελα να πω στη για ερωτήσεις και επεξήγηση. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η δραστηριότητα της αλίας βαθιών υδάτων είναι πρόσφατη. Ήρθε για να καλύψει την ανάγκη έλλειψης ε, άλλων μορφών αλίας και γρήγορα μέσα σε 20 χρόνια οδήγησε σε σημαντικές επιπτώσεις για αυτά τα εκθεία αποθέματα λόγω της πολύ αργής ορίμανσης όπως κατάλαβα. Μιλάμε για ψάρια που αναπαράγεται όπως και οι άνθρωποι αφού ε, φτάσει στην ηλικία των 20. Είναι λοιπόν αργή αναπραγωγή του τους. Το ερώτημά μου είναι πόσα σκάφη στοχεύουν σε αυτού του είδου την αλία. Την αλία βαθέων υδάτων. Τι ποσοστό είναι, είπατε... Ε, μιλάμε για τι ποσοστό του στόλου. Eh, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Εγώ Ευτυχώς ε, μπορώ να μιλήσω με μεγάλη ελευθερία για το θέμα αυτό. Υπάρχουν άλλες χώρες μέλη, των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται περισσότερο όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά όχι η δική μου χώρα. Λοιπόν, καταρχήν, δεν με αφορά αυτό το θέμα. Η Κομισιόν μέχρι τώρα ε, ποτέ δεν έχει κάνει μια παρουσίαση που να μοιάζει με παραμύθι. Και ε, αυτό το οποίο συζητούμε εδώ είναι η απαγόρευση ενός ε, τύπου αλίας που είναι η τράτα. Εάν υπάρχει μια επιστημονική μελέτη σβάφος, η οποία είναι υποεξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν ε, παρέχει καμία επιστημονική αιτιολόγηση για να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ είδα τις συστάσεις που εκδόθηκαν το 2012 για το ίδιο αυτό θέμα, δηλαδή για τα είδη των βαθαίων υδάτων και την αλία στα βαθαία ύδατα καμία από τις ε, συστάσεις δεν σχετίζεται με αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί η πρόταση αυτή προσπαθεί να επιφέρει βελτιώσεις στι τεχνικέ αλίε, να χαρτογραφήσει τον βυθό, να προτείνει κάποια εναλλακτική ε, διαχείριση στις, στα υφαλοπρανή, στα θαλάσσια όρη κλπ. Ε, τώρα, όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων, γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ, όχι σε μια απαγόρευση, για μια απαγόρευση ενός τύπου αλίας, αλλά για μια προστασία και μια ρύθμιση βελτιώνοντας την παρούσα κατάσταση. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, έλαβε υπόψη της ε, τα ΡΑΚ τα οποία αντιβαίνουν στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως λέει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα είδη των ε, βαθέων υδάτων είναι ίσα. Θεωρώ ότι κάτι και δεν ισχύει, γιατί δεν είναι όλα εξίσου ευάλωτα. Το να γενικεύουμε τον τρόπο αυτό ε, μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε περισσότερη σύγχυση και τελικά σαν να δικαιολογήσουμε την πρόταση της κυρίας Επιτρόπου. Τώρα, όσον αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές της ΦΑΟ για τα βαθαία ύδατα, ορισμένες από τις ε, δυνατότητες που απορρίπτει η Επιτροπή θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί ούτω ώστε η πρόταση να μην αποβεί τόσο πολύ εις βάρος ε, του κλάδου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη και πιο επικοδομητική και όχι τόσο επιζήμια για την αλία. Και το κείμενο, για το κείμενο αυτό της Επιτροπής πραγματικά είναι πολύ πιο σκληρό και ριζοσπαστικό από τις ε, δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω σίγουρα να ακούσω τις απαντήσεις της Κομισιόν προς τις ερωτήσεις της κυρίας Φράγκα, οι οποίες ήταν πολύ εύστοχες. Εγώ φυσικά έχω ενδιασμούς για τα βαθιά ύδατα, για τους χαμηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής και η ανησυχία μου είναι ότι μπορεί να προκαλούμε τεράστια ζημιά και ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για την αποκατάσταση αυτή τη ζημιά. Αν κάνουμε κάτι λάθος, λαμβάνουμε υψηλή πίεση από του Γάλλους, ειδικότερα για αυτό το θέμα ίσως να είναι το 1% στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, αλλά ακούω ότι συμμετέχουν κυρίως γαλλικά σκάφη, αν αυτά τα μέτρα ε, όπως ε, έχουν σκοπό θέσουν σε μειονεκτική θέση τους Γάλλους ε, αλείς. Θα ήθελα να υπάρξουν μέτρα που θα υποστηρίξουν τη διαφοροποίηση την μεταφορά του σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αλλά ήθελα να μου πείτε, εάν δεν λάβουμε μέτρα, ποιε θα είναι οι συνέπειε για το θαλάσσιο περιβάλλον, για το μέλλον αυτών των αποθεμάτων και εν τέλει για τους ίδιους τους αλληλείς εάν συνεχίσουμε όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, γιατί μιλάμε για μια τεράστια περιοχή. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πόση ζημιά είναι δυνατόν να κάνουμε ακόμη και αν αυτή η ζημιά κάθε φορά είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αντίθετα από την κυρία Φράγκα, εμείς, ε, εμάς την καλή μας αφορά το θέμα αυτό. Από την άλλη αγαπητέ μου Μπερνάρ, πρέπει να πω ότι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, αλλά εδώ κάνεις τρομερό λάθος έχοντας ακούσει αυτά που λες, τα λέω. Στο άρθρο 9 που προτείνεται, στον κανονισμό που προτείνεται, καταδικάζει η Επιτροπή αυτού του είδους την αλία βαθέων υδάτων και προτείνει την πλήρη κατάργησή της. Νομίζω λοιπόν ότι απευθείας δαιμονοποιεί αυτή την αλία ή την στιγματίζει. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ως εξής μεταξύ επιστημονικών αποδείξεων και γενικοτήτων ε, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα που ασκείται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Σκοτία εξαιτία αυτή τη πρώτη επιτροπή, όπω η Κάρμεν Φράγκα προηγουμένω, η Αλία ε, βαθέων υδάτων στο Κονκαρνό και στην Πουλόνια ασκείται από το 2003. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα διαχείρισης, ποσοστώσης, απαγόρευση αλίευσης κάποιων ειδών, ε, αυστηρά μέτρα εποπτείας, ελέγχου, για, ε, τα αλιεύματα δεν μπορούν να εκφορτώνονται παρά μόνο σε κάποια λιμάνια, παρατηρητές επιτόπου και η διάγνωση που έκανε η επιστήμη το 2012 είπαν ότι αυτού του είδους η αλληλεία γίνεται σε ε, ποσοστό βιώσιμο. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν ε, γίνεται αλίευση με τέτοιου είδους στράτες βυθού, υπάρχει περίπτωση γρήγορα να αποκατασταθούν τα αποθέματα, υπάρχουν νέε καινοτόμε στράτες που χρησιμοποιούνται και το χαιρετίζω, ώστε οι επιπτώσεις να είναι πάρα πολύ περιορισμένες επί του βυθού τη θαλάσση και αυτά που ελέγονταν εδώ και δέκα χρόνια ίσω δεν ισχύουν σήμερα. Η καταστροφή λοιπόν είναι ελάχιστη, χάρη στη δημιουργία κλειστών ε, ε, ζωνών και στο πάγωμα δραστηριοτήτων που επιβάλλουν οι ίδιοι οι αλείς περνούν από μια περιοχή και δεν ξαναπερνούν. Οι ίδιοι λοιπόν περιορίζουν τις ίδιες ε, τις δραστηριότητες και οι απορρίψεις είναι ελάχιστες. Δεν τα λέω εγώ αυτά, οι επιστήμονες το λένε. Και η Επίτροπος πάντα μας λέει εγώ πρέπει να βασίζομαι στα ευρήματα των επιστημόνων. Το ίδιο λέμε και εμεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό μα λένε λοιπόν οι επιστήμονε και οι ερευνητέ. Ότι υπάρξει, είχε υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τι γνώσει που έχουμε για το οικοσύστημα βαθέων υδάτων. Έχουμε χαρτογράφηση, έχουμε έρευνε εκ μέρου ερευνητικών κέντρων. Υπάρχει ένα φάκελο του Ιουλίου του 2012 που λέγει ότι η διαχείριση τη παρούσα αλία ε, σταμάτησε την υπεραλίευση ε, ειδών αλίες βαθέων υδάτων, οι στόχοι για την προστασία των οικοσυστημάτων γίνονται σεβαστοί και το να ε, απαγορευθούν οι τράτες βυθού ή τα στάσιμα απλά διαδίχτυα βυθού είναι κάτι το οποίο στις περιοχές αυτές, Μεχτή, Μπουμπουλόνιο και Κονκαρνό, θα δημιουργήσει πρόβλημα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον έμες σε απασχόληση 600 στην περιοχή. Πιστεύω εγώ ούτως ή άλλως ότι θα πρέπει αυτό το άρθρο 9 να το αναδιατυπώσουμε και να το μελετήσουμε εκ βαθέων, μιλώ για την πρόταση της Επιτροπής, και προτείνω, ο κύριος Αρσένης ήδη το έκανε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, να προτείνουμε εμείς στην Επιτροπή μας να γίνει ακρόαση των ειδικών του κλάδου και των επιστημόνων που θα μας φωτίσουν με συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Συμπερασματικά θα πω ότι μας λέει η Επίτροπος ότι βασίζομαι σε επιστημονικά αποτελέσματα και εμείς λέμε το ίδιο και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σαφή. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πέρα. Ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημαντικές πτυχές. Το, δηλαδή το άρθρο 5, το οποίο ρυθμίζει την πρόσβαση στην ελληνική προσπάθεια και πιστεύω ότι δημιουργεί διακριτική μεταχείριση των χωρών με ποσοστώσεις κάτω των δεκατόνων και τις χώρες ε, που ανταλλάσσουν τις ποσοστώσεις τους. Η άλλη πτυχή είναι το άρθρο 10 ε, εδαφείο Β που αφορά τα σχέδια κλεισίματος των αλληλευτικών ε, περιοχών. αν δεν αλλάξει η αλληλευτική προσπάθεια και αυτό δημιουργεί διακριτική μεταχείριση κατά αλλιέων στη Βορειά Θάλασσα. Αντί να κλείσουμε λοιπόν τους ιχθυότοπους, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ρωτήσει γιατί δεν υπάρχουν ε, επιστημονικά στοιχεία γι' αυτό και σίγουρα να διασφαλίσει οικονομικούς πόρους για τέτοιες μελέτες. Αυτά τα δύο σημεία μου φαίνεται ότι δημιουργούν διακριτική ε, μεταχείριση και ελπίζω ο κ. Αρσένης να τα λάβει υπόψη του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόμας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι Συμμερίζομαι σε όσα χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να βασιστεί πάνω τους βάσει των όσων είπε και ο κ. Αρσένης ότι εδώ μιλάμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά και ότι μιλάμε και για είδη αναπαραγωγική μας εξαιρετικά αρχής και ότι οι συνθήκες εκμετάλλευσης είναι κάτι που προέκυψε πρόσφατα αυτή είναι επαρκής λόγοι ώστε να ε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτού του είδους δραστηριότητε. δραστηριότητες. Και εκτός από προσοχή, το έργο μας πρέπει να βασιστεί σε πραγματικότητες και σε όχι σε... Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σήμερα την Κομισιόν για ποιο λόγο αντί να βασιστεί στις επιστημονικές εκθέσεις βασίζεται σε υποθέσεις. Διότι όπως και να το κάνουμε. Αφενός έχουμε μια επιστημονική έκθεση που κυκλοφόρησε κάποιο καιρό πριν από το σχέδιο κανονισμού της, το οποίο δεν έλαβε καθόλου υπόψη, παρότι αυτό το πρόγραμμα είχε επικυρωθεί από εμάς. Δεν το γνωρίζαμε όλο απαραίτητο καλά. Δεύτερον, η Κομισιόν δεσμεύτηκε ζήτησε για 10 εκατομμύρια ευρώ τρεις μελέτες για τις επιπτώσεις για το βυθό μια μελέτη για τα μέσα περιορισμού των απορρίψεων και των επιπτώσεων ε, στο θαλάσσιο βυθό και μια τρίτη μελέτη είπα, ε, σχεδόν για 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο μέχρι σήμερα καμία από αυτές τις μελέτες δεν έχει κοινοποιηθεί. Δεν έχουμε λοιπόν στα χέρια μας την ε, απαραίτητη βάση για να μπορούμε να συζητήσουμε. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω και να προτείνω είναι να έχουμε στα χέρια μας το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις μελέτες και βάσει αυτών των μελετών να επιχειρηματολογήσουμε. Ελπίζω, δηλαδή δεδομένη τη τιμή που κόστησαν σε δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να μπορούν να αποτέλεσουν τη βάση για να συζητήσουμε. Και συμφωνώ με την πρόταση ή να γίνει κάποια ακρόαση, όσο το δυνατόν πιο ευρεία, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε τους εισηγητές και τους συντάκτες των μελετών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τόμας, ο κύριος Ρομέρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω πλήρως την Επιτροπή της ε, Κομισιόν. Ορισμένοι από εμά περιμέναμε για πολύ καιρό να γίνει κάτι τέτοιο και ε, περιμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί αυτός ο τύπος αλίας. Γιατί απλώς θα τα εναλλακτική. Εάν δεν το κάνουμε με το σωστό τρόπο, η εναλλακτική λύση προκειμένου να εκπληρωθούν κάποια ψηφίσματα των εθνών που ζητούν να υπάρξει μια καλύτερη ρύθμιση και καλύτερη προστασία αυτού του τύπου των οικοτόπων θα είναι το κλείσιμο της Αλίας. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασης αλλά θα πρέπει να ληφθούν πολύ αυστηρά μέτρα ούτω ώστε να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και είναι αναγκαίο να υπάρχουν βεβαίω οι μελέτες αντικτύπου, αλλά θα πρέπει να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση. Έτσι λοιπόν αναμένουμε ανυπόμονα την συνεργασία με τον Κρήτον Αρσένη. Τους έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση από το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οι αλείς κατά πρώτο λόγο και ε, κατά δεύτερο λόγο, εκείνα τα τμήματα του κλάδου προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά του τύπου αλεία. Γνωρίζω ορισμένε ανησυχίε του κλάδου όσον αφορά του κινδύνου ορισμένων ε, τύπων αλίευση με τράτα. Εάν ε, δεν αλλάξουμε δραστικά ορισμένες πρακτικές αλίες, τελικά ε, θα διενιστεί η κατάσταση του παρελθόντος χωρίς να υπάρχουν ξεκάθαρες ε, λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λέβεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν ακούω όλα αυτά τα επιστημονικά πορίσματα τα οποία βλέπω ότι δεν έλαβε υπόψη η Επιτροπή, είδα, ελέγχοντας τη ότι ζητήθηκε από την ΕΑΦ για τον Οκτώβριο του του 2012 μια μελέτη για τα αποθέματα που αφορούν 16 είδη αλλιεύματος. Για κάποια λέγεται ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, για κάποια άλλα ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση των αποθεμάτων κάτω από τα σημεία αναφοράς, για άλλα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε μελέτη, για κάποια άλλα. Τέλο πάντων, αυτά όλα τα και τα σκυλόψερα, τα πορτογαλικά σκυλόψερα, τα σκύμνα σκυλόψερα, ότι δεν υπάρχει ε, στοιχείο Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το α, για το β είδος αλίας. Τελικά δεν μπορεί κανείς για τα αποθέματα να έχει κανένα στοιχείο για τα περισσότερα, για δέκα διαφορετικά είδη τουλάχιστον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εκμετάλλευση όλων αυτών των αποθεμάτων και των ειδών βαθέων υδάτων που ξέρουμε ότι στην ορίμανση φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία αργά και κάποια από αυτά τα νεογνά τους τα φέρουν για περισσότερο από ένα χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτά τα αποθέματα να ζήσουν και να αναπτυχθούν πριν να τα εξαφανίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λέβιν. Κύριος από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα σημεία με το ερώτημα. Για πόσα είδη στοχεύουμε εξαρτάται από τα είδη, διότι βασίζεται ο κανονισμός σε ποσοστά, σε κατόφλια. Πιστεύουμε ότι αναχώρα στην ε, Γαλλία μιλούμε για 30-50 λιευτικά σκάφη, περίπου τα ίδια στην Ισπανία και αυτό που είναι πιο σημαντικό, 30 με 50 είναι ο αριθμός των λιευτικών σκαφών. Αλλά μπορούμε να σας δώσουμε πιο επεξηγηματικά στοιχεία για να είμαστε και πιο ε, ακριβείς. Για να δούμε αν, τι είδους μέσων χρησιμοποιείται, ε, αν έχουμε να κάνουμε με παραγάδια, με τράτες, με δίχτυα βυθού, ποια στιγμή του χρόνου, ποιο χρόνο, με παρασυρώμενα παραγάδια κτλ. Μικρό ε, αριθμό ε, τράτες βυθού έχουμε. Το ανέφερε και ο κύριος Καντέκ και όλα αυτά τα είδη υπάρχουν στον κανονισμό. Τώρα, όσον αφορά τις στράτες και τις στράτες βυθού, τα στοιχεία μπορούμε να σας τα στείλουμε. Έχουμε κάνει μελέτη, έχουμε κάνει μελέτη επιπτώσεων. Η ISIS κάθε δύο χρόνια έως το 2020 μας δίνει κάποια στοιχεία. Όπως είπα, Κάποια τέτοιου είδους αποθέματα έχουν ήδη αλλιευθεί, έχουν γίνει από την ISIS κάποιες συστάσεις. Μπορούμε να καθορίσουμε το επίπεδο βιώσιμης αλίευσης, αλλά κάτι το οποίο βλέπουμε σε αυτά τα οποία λέει ο Σάισις είναι ότι μάσα ε, εφιστά την προσοχή συστηματική ελεία τέτοιων ειδών. Τώρα, γενικά, για να αναφερθώ σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν για τις μελέτες. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο δεν είναι, είναι ακόμη η οι Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία λέγονται. Όπως είπατε, όντως χρηματοδοτήσαμε μελέτες μία από τις οποίες ολοκληρώνεται και θα δημοσιευθεί στο τέλος του παρόντος έτους, έχουμε ζητήσει και αναθέσει ειδικέ μελέτες σε Ινστιτούτα ε, του κλάδου για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αλλιεύοντας με τον πιο ε, βιώσιμο τρόπο και είναι τα πιο ειδικά σκάφη. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αν υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός, κονδύλια από, από το ειδικό ταμείο, ώστε να αλλάξει ο ίδιο, το είδος των αλλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται, να αλλάξουν κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια εργαλεία, κάποιο εξοπλισμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αν δεν πάρουμε μέτρα. Εν μέρη το ξέρουμε, εν μέρη το γνωρούμε. Ξέρουμε ότι οι τράτες μπορεί να είναι καταστροφικές σε κάποιες περιπτώσεις, άρα θα υπάρχει ενδεχόμενα κίνδυνος να καταστρέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Γι' αυτό πρέπει να χειριστούμε και το θέμα των ε, απορρίψεων καθώς και των παρεπιπτών των αλλιευμάτων. γιατί αλλιεύονται καμιά φορά και είδη τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς βρώση και τα οποία πρέπει να ξαναρίχνουμε στη θάλασσα. Και πολλές φορές το ποσοστό τους είναι 50 με 60%. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κανείς αλλιεύσει τέτοιου είδους ε, ε, ε, ψάρια που δεν είναι κατάλληλα προς βρώση, τα ξαναρίχνει πίσω. Ας χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα για να δείτε τι γίνεται να ρυθμιστεί η κατάσταση. Η αλληλευτική προσπάθεια ενός αλληλευτικού στόλου μίας χώρας το 2000 ήταν 30.000 κιλοβατόρες ημερησίως και σε μερικά χρόνια έπεσε σε δέκα χρόνια σε μία, σε χίλια. Χίλιες κιλοβατόρες ανή μέρα. Πρώτα απ' όλα ότι οικονομικά αυτό δεν είναι βιώσιμο και δεύτερον διότι εξαντλούνται σιγά σιγά αυτά τα αποθέματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και τις οικονομικές και τις ε, κοινωνικές επιπτώσεις Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να βρούμε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα, το ποιες είναι οι περιοχές και τα είδη που επηρεάζονται, τι γίνεται από αυτές τις δραστηριότητες. Αν θέλετε όλα αυτά μπορώ να σας τα δείξω, τα συγγεία και να τα συζητήσω. Κάτι όμως το θα ήθελα να πω επί τούτης, είναι ότι το άρθρο 9 του κανονισμού ασχολείται με ειδικέ τεχνικές ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστά αυτή την δραστηριότητα και η ελευτική στόλη των ε, Ισπανών και των Πορτογαλών ε, με τα παρασυρώμενα παραγάλια δεν καλύπτουν αυτόν τον κανονισμό. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω εξήγηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αμέσως μετά από αυτό που είπατε σηκώνονται χέρια. Ο κύριος Αρσένης πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ακρόαση. Θα πρέπει οι συντονιστές να αποφασίσουν για μια ακρόαση και πιστεύω ότι θα αποφασίσετε για τον Ιανουάριο. Το δεύτερο, αυτό που καθίσατε σαφέ μετά από τις διευκρινήσεις της Κομισιόν, είναι ότι το όλο θέμα δεν αφορά απαγόρευση της αλίας ε, στα βαθιά νερά. Είναι απαγόρευση των μη επιλεκτικών μέσων, όπως είναι οι τράτες βυθού. Όπως κατάλαβα, υπάρχουν άλλες χώρες Άλλε χώρε που το χρησιμοποιούν και άλλε χώρε που δεν το χρησιμοποιούν. Άλλε χώρε χρησιμοποιούν παραγαδιάρικα που δεν θα απογορευτούν σε, σε καμία χώρα και που είναι πιο επιλεκτικές ε, ως μέσα. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερα ε, στοιχεία για αυτά. Δεν ήταν σαφές. Είπατε περίπου 30 με 50 σκάφη αναχώρα αλλιεύουν σε βαθέα ύδατα. Αλλά είπατε κάτι άλλο για τη Γαλλία, δύο ή τρία. Μπορείτε να μας δώσετε καλύτερα, πιο, περισσότερα στοιχεία, ποια πλοία θα, ποια θα επηρεαστούν από αυτή την νομοθεσία. Διότι όπως κατάλαβα δεν μιλάμε για αλληλεία σε βαθιά δεν μιλάμε για τις στράτες βυθού που στοχεύει αυτός ο κανονισμός. Ε, και εμένα η ερώτησή μου αφορά το ίδιο θέμα. Αν μιλάμε για δύο-τρεις στράτες βυθού, μιλάμε για μια τεράστια περιοχή. Γιατί τόσο λίγα σκάφη. Δεν ξέρω καλά το σύστημα των ποσοστώσεων. Υπάρχει κάποιο περιορισμό. Ή... Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούνται οι οικονομικές δυνατότητες εφόσον υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Σενιόρ Καδέκ. Ο κ. Καδέκ. Μια μικρή παρατήρηση για την Κομισιόν. Ο κύριος Αλαβιζό που είναι γνωστός επιστήμονας ε, και αναγνωρισμένος ε, μιλάει για υπερβολές και παραπληροφόρηση. Θα ήθελα λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά διότι δεν έχω συνηθίσει να μην πιστεύω τον κύριο Λαμπιζό που είναι τόσο αξιόπιστος και γνωρίζει καλά τη δουλειά του. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, να μας δοθούν καλύτερες πληροφορίες. Καλό είναι λοιπόν που ζητείτε αυτή η ακρόαση, είναι απολύτως απαραίτητη. Επίσης, ε, το προλαμβάνω, μιλάμε για μια μορφή αλίας εξαιρετικά ρυθμιζόμενη. Στη γαλλικά λέμε ζώνη και τυράντες. Ε, υπάρχουν ε, κλειστές περιοχές, συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα, δορυφορική παρακολούθηση, παρατηρητές επί των σκαφών. Τι άλλο να κάνουμε όταν οι ίδιοι επιστήμονες μας λένε ότι τα είδη δεν βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι όλα τηρούνται. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την πρόταση τη ε, ε, ε, της Επιτρόπου, η οποία πάντα μα λέει ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικέ γνωμοδοτήσεις. Κύριε Στόμα. Oui, Κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που επιτέλους είπε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πρόκειται πράγματι για τις στράτες βυθού που στοχεύονται εδώ και που απαγορεύονται γίνονται αντικείμενα απαγόρευση. Άρα λοιπόν βρίσκω κάπω παράδοξο το γεγονό ότι καταρχήν μα εξήγησαν ότι επιλούνται τα είδη και ε, για να μας πούν κάτι άλλο στη συνέχεια. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την απαιτούμενη επιστημονική αυστηρότητα την οποία ε, θα στην οποία θα πρέπει να περιοριστούμε την οποία θα πρέπει να τηρήσουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια έρευνα η οποία ε, στήχησε πάνω από 3 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία στοχεύει το ζήτημα του αντικτύπου στα ε, οικοσυστήματα μεγάλου βάθους και επίσης υπάρχει μία έρευνα όσον αφορά τις απορρίψεις και νομίζω ότι αυτή στήχησε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ Άρα λοιπόν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτές τις έρευνες ούτως ώστε να μπορέσουμε με κάθε επιστημονική αυστηρότητα να, και πολιτική αυστηρότητα να αποφασίσουμε. Και αν ε, η πρόταση του εισηγητού του κ. Αρσένη είναι να γίνει μια ακρόαση τον Ιανουάριο, ε, θα ήθελα να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις έρευνες αυτές μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ε, πράγματι θα θέσουμε στη διάθεσή σας τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ε, τον αριθμό των ε, σκαφών που επηρεάζονται από τον κανονισμό αυτό. Για να επανέλθω στο θέμα αυτό των δύο ή τριών σκαφών. Έθεσα απλώς το παράδειγμα της γαλλικής αλίας βαθέων υδάτων και τα πράγματα υφροπούνται από χώρα σε χώρα βεβαίως. Αλλά αν πάρουμε τη Γαλλία υπάρχουν δύο μεγάλα σκάφη αλίας βαθέων υδάτων που στοχεύουν ακριβώς αυτά τα είδη και χρησιμοποιούν την τεχνική της στράτας. Υπάρχουν άλλα σκάφη που ε, αλλιεύουν αλλιεύματα ε, βαθέων υδάτων και τα οποία εν μέρει απορρίπτονται. Ο κανονισμός έχει σαν σκοπό να ρυθμίσει μέσω ορισμού ενός κατοφλίου, ενός ποσοστού δηλαδή αλλιευμάτων και ένα κατόφλι του βάρους, εκείνα ε, στα οποία στοχεύει, αποσκοπεί ο κανονισμός. Ούτως ώστε να ελεγχθούν οι επιπτώσεις στα βαθέα ύδατα, στα αποθέματα των βαθέων υδάτων. Ε, υπάρχει ένα κάπως ασθενές ε, όριο όσον αφορά τα λεύματα βαθέων υδάτων. Θα πρέπει να οριστεί ένα συγκεκριμένο κατόφλι το οποίο να αφορά τα λεύματα των βαθέων υδάτων και να μην ε, αφορά τα άλλα λευτικά σκάφη τα οποία ασκούν τη συνήθεια λευτική τους δραστηριότητα και λέγουν και κάποια είδη τα οποία δεν θεωρούνται ότι είναι βαθέων υδάτων. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, θα υπάρξουν εκείνα τα οποία καλύπτονται, τα είδη αλευμάτων, βαθέων υδάτων, τα οποία καλύπτονται αυτόν τον οργανισμό και αυτά τα οποία δεν καλύπτουν. Θα υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, το πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυριπάτη. Ε, και στο θέμα αυτό θα ακούσουμε καταρχήν την παρουσίαση αυτού του νέου πρωτοκόλλου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχήν. Εκ μέρους της Επιτροπής έχει το λόγο ο κύριος Πέγκ. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το νέο πρωτόκολλο για την αλληλεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρίμπατη. Θα υπενθυμίσω κάποια στοιχεία για τη δημοκρατία του Κυρίμπατη που βρίσκεται στον Ειρηνικό, που έχει... Που έχει τη μεγαλύτερη ΕΟΖ. Ελάχιστοι κάτοικοι, 5.000. Πρώτη οικονομική δραστηριότητα είναι η αλληλεία. 80% είναι αλληλείς. Σε αυτή την ΑΟΖ έχουμε πάρα πολλούς αλληλευτικούς στόχους από την Κίνα, την Ταϊβάν, την Κορέα και την Αμερική. Όσον αφορά την παρουσία ε, του Ευρωπαϊκού Αλευτικού Στόλου είναι περιορισμένης εμβέλειας, δηλαδή περίπου τέσσερα γρήγοροι και οι δυνατότητες αλίευσης στο δυτικό και κεντρικό μέρος του Ειρηνικού είναι πάρα πολύ περιορισμένοι, δεδομένου ότι τα αλιευτικά μας σκάφη αλλιεύουν το 2-3% των αλλιευμάτων στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τον αλλιευτικό μα τόλο και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η συμφωνία, δεδομένου ότι για τον αλλιευτικό μα τόλο το γεγονός ότι έχει δυνατότητα αλλίε στον ειρηνικό εξασφαλίζει παρουσία και ε, στοιχεία ε, που αφορούν ε, μία τόσο σημαντική δραστηριότητα και για μας σημαντικού και για την Λατινική Αμερική. Πιστεύω ότι την ε, συμφωνία του Κυρίμπατη θα πρέπει να τη δούμε ως κάτι το σημαντικό σαν αφορά την πολιτική διάσταση του όλου θέματος. Χάρη σε αυτή τη συμφωνία μπορούμε να έχουμε μια κάποια βαρύτητα και να μπορέσουμε να περασπιστούμε τις αρχές της ε, ε, αηφορίας στην περιοχή αυτή. Με τις παρούσες δυσκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή με τα πρωτόκολλα, δηλαδή με την Μικρονησία και τα νησιά Σαλομών, είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει αυτή η συμφωνία και το πρωτόκολλο εκεί με την ε, δημοκρατία του Κυρίμπατη. Φάνω τώρα στα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά αν θέλετε αυτής της συμφωνίας που στις 3 Ιουνίου έχει τριετή ισχύ και θα καλύψει τις δραστηριότητες του ελευτικού μας στόχου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Η δική μας ε, χρηματική ε, συνεισφορά είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, 350 δις, 350 εκατομμύρια δίδονται στην υποστήριξη του κλάδου αυτού και την διαχείριση της αλίας στην Δημοκρατία του Κυρίμπατη και συμπεριλαμβάνεται εδώ και η ανάπτυξη των έργων υποδομής και η κατάρτιση και ο έλεγχος και η εποπτεία της αλίας σε αυτή την ΟΣ. Τώρα, όσον αφορά την χορηκτικότητα αναφοράς, που χαρακτηρίζει το νέο πρωτόκολλο είναι 15.000 τόνοι ετησίως. Πρόκειται για χωρητικότητα αναφοράς που λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και λαμβάνει συγχρόνως υπόψη το επίπεδο των αλλιευμάτων έτσι όπως ε, είχαν προβληθεί στο προηγούμενο πρωτόκολλο που είχαμε 6.400 τόνους, αλλά de facto αλλιεύουμε πολύ περισσότερο, διότι κατά μέσον όρο αλλιεύουμε 12.000 τόνους. Οπότε λοιπόν, αυτός ο αριθμός αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, διότι είχαμε ξεπεράσει 13.000 τόνους το 2011. Τελικά λοιπόν πρέπει να πω ότι η χωρητικότητα ε, αναφοράς αφορά τους πραγματικά αλλιευόμενους τόνους. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στην Γαλλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία να έχουν αλλιευτικά σκάφη. Έχουμε τέσσερα αλλιευτικά σκάφη με παραγάδια και τέσσερα, τέσσερα πέντε γρηγροί από αυτές τις ε, χώρες. Οι εφοπλιστές έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια στον τομέα αυτό, διότι έχουν καταβάλει άνα σκάφος 300.000 ευρώ για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα του Κυρίμπατη. Η άλλη οικονομική συνεισφορά που καταβάλλεται από άλλους είναι επίσης σημαντική. Έχουμε οικονομική συνεισφορά στο Ταμείο Παρακολούθησης, πράγμα που μας υποχρεώνει ε, ε, η συμφωνία με την παρουσία παρατηρητή και άλλες δαπάνες επίσης για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία είναι σημαντικές και τις απομίζονται υπεύθυνοι. Υπάρχει, όπως ξέρετε, συζήτηση όσον αφορά το ΒΕΝΤΕΣ. Στην αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης, το κυρίμπατη ήθελε να έχει το VDS. Εμείς ζητήσαμε να μην υπάρχουν, διότι το επιθυμούσαν και τα κράτη-μέλη και ο ελευτικός στόλος, αλλά υπήρξε δυσκολία στη διαπραγμάτευση και ότι θα πρέπει να πληρώσουμε κάποιο τίμημα για να έχουμε αυτή τη συμφωνία με το κύριο Μπατή. Αλλά δεδομένου ότι είναι κάτι που είναι σημαντικό για τον ελευτικό μας ε, στόλο, θα θέλαμε να συνενέσει για να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή, το κοινοβούλιο, στην καταβολή αυτού του ποσού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα δίδω το λόγο στην κυρία Λόβιν, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Κατά βάση λοιπόν, εάν ε, διαβάσουμε την αξιολόγηση, μία από τις ε, συστάσεις που προκύπτουν από την αξιολόγηση είναι ότι θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης για τα αλευτικά μέσα. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλου μεγέθους ε, τόνοι ως παρεπίμπτοντα αλλιεύματα με αυτόν τον τύπο αλλιεύσης. Ε, υπάρχει περιαλίευση των θηνοειδών μια μείωση της ε, θνησιμότητας κατά 80% έστω και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μικρό μερίδιο των συνολικών αλλιευμάτων θηνοειδών στην περιοχή αυτή παρόλα αυτά σύμφωνα με την αξιολόγηση ε, θα έχει ε, αυτό ένα σημαντικό αντίκτυπο στην θνησιμότητα αυτού του είδους τόνου. Και πέρα από αυτό υπάρχουν παρεπίπτοντα αλλιεύματα καρχαριοειδών περίπου 48 ε, και 80 χιλιάδες καρχαριοειδή ω ως παρεπίπτοντα αλεύματα ε, ε, ήδη περιλαμβάνονται μεταξύ των επαπειλούμενων ειδών. Για να μειωθούν λοιπόν τα παρεπίπτοντα αλεύματα των καρχαριοειδών και των νεογνών των θηνοειδών θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα διαχείρισης το οποίο να βασίζεται στη μελέτη αξιολόγηση. Και δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο στην συμφωνία. Ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να μας, να μας πει κάποια περισσότερα πράγματα σχέση με αυτό. Όσον αφορά την αξιολόγηση, είπατε ότι υπάρχουν τρεις χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, θα αξιοποιήσουν αυτές τις λευτικές ευκαιρίες. Ε, έξι γρηγροί, ε, τράτησαν με σιρτή. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το πρωτόκολλο προβλέπει 12 τράτες με σιρτή που δεν αξιοποιούνται. Άρα η αξιοποίηση είναι 0%. Ενώ η σύσταση λέει ότι εφόσον δεν αξιοποιηθούν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να δούμε τι γίνεται με αυτή την αξιοποίηση των γρηγρή. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να γίνει διαπραγμάτευση σε σχέση με το θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση αποθεμάτων, ε, εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ε, υπεραλίευση ορισμένα είδη, αλλά για το κίτρινο τόνο εδώ συντρέχει κίνδυνος υπεραλίευσης και τα ποστά θνησιμότητας θα πρέπει να μειωθούν εδώ. Έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο και θα ήθελα να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα εν σχέση με το πώς προτίθεστε να πετύχετε κάτι τέτοιο. Και διερωτώ με ε, ε, ε, το εξής, η Επιτροπή μετέφερε, ανέφερε αυτό το μοντέλο, περιφερειακό μοντέλο αλίευσης. Ξέρετε, δεν υπάρχει πρωτόκολλο στη Μικρονησία, γιατί ε, δεν ήθελα να, γίνει το πρωτόκολλο χωρίς ε, να συμπεριληφθεί αυτό το ημερήσιο μοντέλο. αυτό το μοντέλο. Η Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί μια συμφωνία για 50.000 τόνους. Αλλά το πρωτόκολλο επίσης δέχεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετα αλλιεύματα, άρα δεν υπάρχει ένα ανώτερο κατόφλι όσον αφορά τις αλληλευτικές δυνατότητες εδώ. Και πώς όλα αυτά ε, συμφωνούν με τη μείωση της ε, θνησιμότητας των αλλιευμάτων σε αυτή την περιοχή. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της αναπτυξιακής βοήθειας. Η Επιτροπή αναφέρει ότι ένα ουσιαστικό τμήμα αυτού του ελευτικού πρωτοκόλλου είναι η εταιρική σχέση, η οποία θα οδηγήσει σε μια στήριξη του κλάδου. 350.000 ε, ευρώ. Αλλά όταν διαβάζω την ε, αξιολόγηση με καταπλήσει το γεγονό ότι όταν ε, βλέπουμε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και τα έγγραφα για τη στρατηγική της χώρας, για την περιοχή αυτή, δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα από το EDF που να πηγαίνει στους αλείς. Παρόλο που το 10ο πρόγραμμα EDF ε, περιγράφει λεπτομεριακά στο στρατηγικό του κείμενο ότι η διαχείριση των εθνικών πόρων αποτελεί μία από τις προτεραιότητές τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί κατ' ουσία 13 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα ληφτικά προγράμματα στην περιοχή αυτή. Αλλά το Κυριμπάτι ε, μέχρι στιγμής ε, δεν ήταν επιλέξιμο ε, για αυτού του είδους τα προγράμματα. Γιατί έχουμε ένα FPA όσον αφορά το Κυριμπάτι. Άρα λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα επωφελούνται από την τομεακή υποστήριξη. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να μας απαντήσει σχετικά η Επιτροπή, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Κυριμπάτι έχασε την ευκαιρία να λάβει η DF στον αλληλευτικό τομέα στη βάση των διαφόρων προγραμμάτων, λόγω ακριβώς του FPA. Ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα σε σχέση με το πώς έχει ακριβώς χρησιμοποιήσει την ε, τομεακή υποστήριξη στο παρελθόν και ποια ήταν η αποτελεσματικότητά της. Και θα ήθελα να επιθυμίσω στους συναδέλφους ότι το Κυριμπάτι είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα σε αυτή την περιοχή. Και η δεύτερη τα, τα, τα, τα, τα, σε δεύτερη σειρά πιο σημαντικά έσοδα για τη χώρα προέρχονται από την αλία. Εάν θέλουμε λοιπόν να, παρέχουμε, να παράσουμε αρτισακή βοήθεια στη χώρα αυτή, ε, θα πρέπει να δοθεί στην ε, γεωργία και στην αλία, που είναι η βασικότερη κλάδη. Αλλά θα έπρεπε να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φράγα. Sí. Tenía pedida la palabra, la tenía apuntada. No, no. Κάποιον άλλο άκουσα, δεν άκουσα το όνομά μου. Μπάς περιπτώσει. Άκουσα την Επιτροπή. Νομίζω ότι κατόρθωσε να κάνει συμφωνία με το Ρίμπατη, που είναι η μοναδική συμφωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή με τον Ειρηνικό και κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα κοινοτικά των αλλιευτικά σκάφη μας. Τέσσερα σκάφη δηλαδή. Για αυτά μιλάμε. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάποια από τα θέματα που έθεσε η κυρία Λέβιν είναι σημαντικά και αφορούν την επιστημονική επιτροπή την ειδική που υπάρχει που λειτουργεί όπως λειτουργεί εν περιπτώσει. Τώρα όσον αφορά το σύστημα του Vessel Day Scheme λειτουργεί και αυτό όπως λειτουργεί δέχεται κάποιες χώρες και εφαρμόζεται βασικά αυτό για να βάλει λεφτά στην ταμεία του. Το Day Vessel Skin αφορά, δεν αφορά ούτε τα εγχώρια αλλιευτικά σκάφη, ούτε αυτά τα οποία δραστηριοποιούνται με την βενθαπελαγική ε, αλληγία αλία. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο είναι αδιαφανές, αλλά τι να γίνει. Τέλος πάντων, εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο με αφορά στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, όχι μόνο αυξάνεται το τίμημα που καταβάλουν οι εφοπλιστές, αλλά δημιουργούνται και νέοι φόροι του οποίους πρέπει να καταβάλουν, όπως λέει και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Το άρθρο 3.4 γίνεται λόγος για 300.000 ευρώ που πρέπει να καταβάλουν τα τον αλλιευτικά για να μπορέσουν να αλλιεύουν κοντά στις παράκριες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι τριπλασιάστηκαν οι δαπάνες που κατέβαλαν και οι τέτραπλασιάστηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι αν το δέχεται ο, κλάδος σημαίνει ότι μπορεί να τα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Τώρα, το άρθρο 12, όπου γίνεται λόγος για ρήτα αναθεώρησης, βλέπω για πρώτη φορά κάτι το οποίο με καταπλήσει. Λέει τα εξή. Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής αυτού του πρωτοκόλου θα αναθεωρηθεί ε, το μέρος που αφορά τον πλειοκτήτη για να μπορέσουν ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Πρώτη φορά βλέπω ότι θα αναθεωρηθεί σε δύο χρόνια το κομμάτι που αφορά τις οικονομικές ε, υποχρεώσεις του πλειοκτήτη ή εφοπλιστή. Τι σημαίνει αυτό μονομερός, διότι εγώ αν μπορέσω να το συγκρίνω με τη συμφωνία που έχουμε για την Γρυλανδία, στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι καταβάλλονται συμβολικά ποσά, δεν υπάρχει αύξηση σε αυτό που ζητείτε να καταβάλουν οι πλειοκτήτες, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη αυτό το οποίο συνεισφέρει ε, το, το ποσοστό με το οποίο οικονομικά συνεισφέρει ο πλειοκτήτης είναι 10%, ενώ εδώ ξεπερνάει το ποσοστό του 40%. Και συνεχίζονται οι αυξήσεις και προβλέπονται και αναθεωρήσεις. Ας μου εξηγήσει η Επιτροπή ποιο είναι το κριτήριό της για τέτοιου συμφωνίε. Γιατί κάποια στιγμή λέμε αχ οι κακόμοιροι δεν έχουν λεφτά και σε άλλου ζητείτε πολύ περισσότερο χρήμα και συνέχεια ε, φευρίσκονται και νέε ρήτρε αναθεώρηση και λέει ότι θα υπάρξει αναθεώρηση μετά από δύο χρόνια εφαρμογή. Βάσει ποιου κριτηρίου. Διότι ή θα πρέπει όλοι να πληρώνουν βάσει των ιδίων κριτηρίων και όχι βάσει του εσύ το Α, εγώ το Β και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανέφερα και πάλι τη Γρυλανδία για να καταλάβει η Επιτροπή. Α μου εξηγήσει λοιπόν αυτή η Επιτροπή περί τίνο πρόκειται. Γιατί για κάποιε συμφωνίε ισχύουν κάποιε αυξήσει, για άλλου όχι. Το θέμα τη Γρυλανδία, που τώρα μόλι αναθεωρήθηκε η συμφωνία τη, δεν δουλεύει έτσι. Α το, μου το πει λοιπόν αυτό η Επιτροπή. Επίση, το άρθρο 12, αυτό το οποίο είναι καινοτόμο και το εφαρμόζει για πρώτη φορά η Επιτροπή, τι ακριβώ σημαίνει. Κανένα άλλο δεν βλέπω να το λόγο. Η Επιτροπή. Α, όχι, και ο κύριο Γκάλαχερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκτός μικροφώνου μιλητής. Το Κυριμπάτι είναι πολύ μακριά από την Ιρλανδία. Αλλά από ό,τι μου λένε είναι ένα πανέμορφο μέρος. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως εμένα είναι όπως θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίασή της και τις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε 15.000 τόνους, δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά, από 80.000. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που από 80 τόσο 15.000 τόνους υπάρχουν στοιχεία επιστημονικά που δικαιολογούν μια τόσο σημαντική αύξηση. Μετά υπάρχουν ε, τέσσερις, ε, έξι ε, γρηγροί και περισσό... και τέσσερα με παραγάδια. Τέλος, αυτό που ήθελα να πω, όσον αφορά τα 300.000 ανασκάφους, δεν έχω ιδέα κατά πόσο αυτό είναι σημαντικό ή όχι, αλλά η αρχή είναι σημαντική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για... Θα μπορούσαμε να, παρέχουμε παρατηρητές επί των σκαφών. Να Πως Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα απαντήσω εγώ με τη σειρά των ερωτήσεων. Θα ξεκινήσω από τη συγκέντρωση των ψαριών είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο των συμφερόντων και των πρακτικών των στόλων που δρούν στις περιοχές. Είναι φυσιολογικό λοιπόν εδώ να μην έχουμε διατάξεις σε σχέση με αυτές τις διατάξεις σε ένα ξεχωριστό παράλογο. Στο πλαίσιο της WCPFC θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, τώρα έχουμε το θέμα του τόνου όπως είπαμε για τον το μεγαλόφθαλμο τόνο και, αλλά αυτός εκπροσωπεί μόνο το 2% των αλλιευμάτων του κοινοτικού στόλου στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Ο κοινοτικός στόλος δηλαδή Δηλαδή μιλάμε για το 2% του 2% διότι ο ευρωπαϊκός στόλος αλλιεύει το 2% μόνο. Πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι το διακύβευμα είναι λίγο σχετικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τα παρακαδιάρικα, το γεγονό ότι περάσαμε από 12 σε 6, λάβαμε υπόψη ένα ποσοστό χρήση μηδενικό στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Διατηρήσαμε μια σειρά αλληλευτικών δυνατοτήτων μετά από αιτήματα από τα κράτη-μέλη και τους τόλους που μας επιβεβαίωσαν ότι μας συμφέρει να διατηρήσουμε αυτού του είδους την αλία στο μελλοντικό πρωτόκολλο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον αυτό που είναι σαφέ, είναι ότι η αξία του πρωτοκόλλου εξαρτάται ελάχιστα από τον αριθμό παραγαδιάρικων που έχουν γραφεί Η αξία είναι ουσιαστικά τα γρήγορα Είναι αρκετά σαφές. Τώρα έρχομαι στην ερώτηση που αφορά την κατάσταση των αποθεμάτων και εκεί να υπενθυμίσω το 80% των αλλιευμάτων του κοινοτικού στόλου είναι λιστάω. Όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι αυτού του είδους τον τόνο, το skipjack, δεν υπάρχει κίνδυνος ε, υπερεκμετάλλευσης, λακέρδας δηλαδή, παλαμίδας. Για τον κυτρινόπτερο τόνο, εκεί υπάρχουν στοιχεία που καταδείχνουν ευαισθησία ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται εξισορρόψη της βιομάζας τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς σε αυτή την κατηγορία τόνου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εκεί πιστεύω επίσης επιβάλλεται και προσοχή σε περιφερειακό επίπεδο δεδομένων των ελάχιστων επιπτώσεων των αλλιευμάτων του Ευρωπαϊκού Στόλου. Όσον αφορά τα επιπρόσθετα αλλιεύματα, θεωρητικά ίσως να μην υπάρχουν όρια όσον αφορά το επίπεδο επιπρόσθετων ελευμάτων στο Κυριμπάτι. Τώρα πιστεύω ότι με τέσσερα σκάφη ο κίνδυνος υπέρβασης είναι σχετικά χαμηλός. Παρατηρούνται ιστορικές τάσεις ε, και έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο περιθώριο. Ο μέσος όρος ήταν 12.000 τόνοι. Έχουμε πάρει ως αναφορά το 15.000 τόνους ως σημείο αναφοράς. Ε, και αυτό είναι ένα περιθώριο που μας επιτρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε υπέρβαση και για τις τρίτες χώρες. Αποτελεί διασφάλιση. Τους λέμε ουσιαστικά ότι αν κατά λάθο υπερβούμε αυτό το σημείο, το επίπεδο αναφοράς, θα καταβάλουμε κάποια πληρωμή για τα αντίστοιχα λιεύματα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αλληλευτικού τομέα στην περιοχή, στο Κυριμπάτι, Πρέπει να υπενθυμίσουμε, πιστεύω, ότι κάθε κράτος επιλέγει τις προτεραιότητες του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, το Κυριμπάτη έχει την επιλογή να εγγράψει την αλία ή όχι μεταξύ των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης. Ε, για τη χρηματοδότηση που λαμβάνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι φυσικά ένα από τα περιφερειακά έργα που έχει αποτελέσματα και που επηρεάζει την κατάσταση του Κυριμπάτη. Ας μην ξεχνάμε επίσης και το εκτακτό τέλος που πληρώνουν οι πλειοκτήτες, στο οποίο σχετίζεται με την επιλογή των πλειοκτήτων να, να αναπτύσσουν την φυσική τους παρουσία, την, ε, το logistics τους ε, στο αρχιπαλαγός του Κυριμπάτη, στα νησιά των Χριστουγέννων, για παράδειγμα, όπου βρίσκονται την εξέλιξη διάφορα αναπτυξιακά έργα, τόσο όσον αφορά τη βιομηχανία εκφόρτωσης και μεταποίησης. και αυτή η τομεατική στήριξη θα βοηθήσει στην υποστήριξη της ανάπτυξης αυτών των έργων που ε, βοηθούν την τοπική οικονομία του Κυριμπάτη. για τα όσα είπε η κυρία Φράγκα. Ναι, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Έχουμε διάφορες ε, αυξήσεις φόρων ή τελών ε, υπερβολικές. Αυτό το έχει δεχθεί ο τομέας. Δεν θα το έλεγα ότι το δέχτηκε ευχάριστα, αλλά ε, γενικά υπάρχουν συμφωνίες που έχουν προτεραιότητα για μας και για τους τόλους και άλλες συμφωνίες που έχουν μικρότερη προτεραιότητα. Το Κυριμπάτι είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Γι' αυτό το λόγο ο Στόλος αποφάσισε να επενδύσει και να παρέχει μια τέτοια χρηματική συμβολή σε αυτή τη συμφωνία. Είναι σαφές ε, ότι αυτός ο κατεξαίρεση χειρισμός του στόλου δεν μπορεί να αναπαραχθεί και στις υπόλοιπες συμφωνίες ε, αλληλείας. Στο άρθρο 2 προβλέπεται αναθεώρηση αυτή τη συμβολή των πλειοκτητών. Αυτή τη ρήτρα τη ζήτησε το Κυριμπάτη στι διαπραγματεύσει. Είναι μια ε, ρήτρα που δεν θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα για να αυξηθεί η συμβολή των εφοπλιστών, αλλά είναι μια απέτηση που χρειάστηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Μιλήσατε επίσης ε, για τις συμβολές και για το ποσοστά που διαφέρουν από συμφωνία σε συμφωνία. Ναι, ισχύει, υπάρχουν σχέσεις ε, ισχύω που διαφέρουν στις σχέσεις μας με την κάθε χώρα. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες που έχουν προτεραιότητα και άλλες λιγότερα. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες για τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι απάντησα σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Το πρόβλημα των παρατηρητών επεκτάθηκε ως το ζήτημα των παρατηρητών επεκτάθηκε ώστε να γίνεται συστηματικά και όσον αφορά τον κοινοτικό προπολογισμό αυξάνεται, αλλά φυσικά ανάλογα με το Άζα αναφορά, το οποίο επίση ευξήθηκε σημαντικά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Φράγκα. Για μια στιγμούλα. Ίσως δεν έκανα με σαφήνεια την ερώτησή μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι οι πλειοκτήτες πρέπει όλο και περισσότερο συμμετέχουν στο συνολικό κόστος της Συμφωνία. Αυτό δεν είχε κάνει τίποτε με την ε, γενικότερη διαπραγμάτευση που αφορά τη σύναψη μια συμφωνίας αληφτική. Όσον αφορά όμως την οικονομική συμμετοχή του πλειοκτήτου και η αύξηση ισχύει για κάποιες συμφωνίες και όχι για άλλες. Και ανέφερα προηγουμένως την Γρυλανδία. Και εγώ ερωτώ. Γιατί αυτό συμβαίνει, ισχύει για κάποιες συμφωνίες και όχι για κάποιες άλλες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μία διαπραγμάτευση που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη χώρα. Αλλά το θέμα της οικονομικής συνεισφοράς των πλειοκτητών και την ε, ε, διαφορετική συμμετοχή τους, ε, τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μου το εξηγήσει. Βάσει ποιας γενικής γραμμής πλεύσεως επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κούρν. Εγώ ήμουνα σκιώδης για την ε, συμφωνία με την Γλανδία και κατ' ουσία είχα θέσει το ίδιο ερώτημα προς την Επιτροπή όπως η Κάρμαν Φράγκα γιατί η νέα συμφωνία την οποία διπραγματευθήκαμε, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσχώρηση της ε, Γρυλανδίας αφορά ένα υψηλότερο τέλος, ενώ το ποσοστό ελευμάτων ήταν ε, μικρότερο από ό,τι στο παρελθόν και είχε αυξηθεί και η συμβολή των ε, πλειοκτητών. Και η απάντηση ήταν ε, ότι αυτό το διαπραγματεύαμε με τους πλειοκτήτες, καθώς και την ποιότητα και τους τύπους των αλλιευμάτων, οι οποίοι είναι εμπορεύσιμοι καλύτερα με τον τρόπο αυτό στην αγορά. Αυτή την απάντηση μου δώσανε. Γι' αυτό έτσι λοιπόν η Γρυλανδία είναι το υπόδειγμα για χαμηλές ε, τιμές. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι η αναμενόμενη τιμή εκφόρτωσης του, των αλευμάτων των 50.000 ε, τόνων στην περιοχή αυτή. Στα προηγούμενα πρωτόκολλα ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος ε, Μπέρκ. Sur Όσον αφορά την εκφόρτωση, την ε, αξία της, δεν έχω κάποια εκτίμηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ε, ξεκάθαρα στοιχεία. Ε, μπορούμε να δούμε ποια είναι η τιμή πώληση κλπ. Αλλά δεν έχω συγκεκριμένου αριθμού να σα αναφέρω σήμερα. Ξέρω ότι η προηγούμενη έκθεση επενέθηκε ω ε, περιλαμβάνοντα μια πολύ καλή σχέση τιμή ε, κόστου ωφέλεια. Και υποθέτω ότι θα πρέπει να ισχύσει και στο επόμενο πρωτόκολλο αυτή η θετική σχέση τιμή ωφέλεια. Όσον αφορά τη συμβολή των πλειοκτητών, η γραμμή που όρισε η ανακοίνωση για τι εξωτερικέ διαστάσει είναι πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή, η συμβολή των πλειοκτητών θα πρέπει να αυξηθεί σε ένα σύνολο πρωτοκόλλων, είτε στον βορρά είτε στον νότο. Δεν ξέρω τώρα, δεν θα σα πω τι ε, λεπτομέρειε τη κάθε διαπραγμάτευση που έγινε με τη Γλανδία, αλλά κάθε φορά πρόκειται για μια ε, πολιτική επιλογή τη ε, επιτροπή που, για την οποία έχει κάποια επιχειρήματα η Επίτροπος ε, και την οποία θα ξαναδούμε στο, μελλοντικά στο σύνολο των ε, αλευτικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Αύριο στις 9 ακριβώς θα αρχίσουμε με την συνάντηση των συντονιστών. Γεια σας, καλό βράδυ και τα λέμε αύριο.